Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους να φύγουν ε, από εδώ μπροστά μετά από τα δύο πρώτα λεπτά όπου τους επιτρέπουμε να πάρουν κάποιες φωτογραφίες του υποψήφιου επίτροπου αλλά μετά τα δύο πρώτα λεπτά παρακαλώ θα πρέπει να φύγετε από εδώ μπροστά μας, να φύγετε από αυτές τις θέσεις. Δύο ανακοινώσει πριν να καλωσορίσω τον ε, προσκεκλημένο μας. Θα ήθελα να ζητήσω από όσου παρακολουθούν ε, την ακρόαση να μην ε, κρατούν θέσεις που σαφώς φέρουν ονόματα άλλων και να σημειώσω ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει από το Γιάν 4Q1, την αίθουσα όπου μεταδίδεται η συζήτηση και επειδή υπήρξαν χειροκροτήματα στη διάρκεια κάποιων ακροάσεων, να θυμίσω ότι μόνο τα μέλη μπορούν να χειροκροτούν εάν το επιθυμούν. Mrs. and me uh, will co-chair uh, Και τώρα η κυρία Λουγκούσκοκ και εγώ θα συμπροεδρεύσουμε σύμφωνα με τη διαδικασία και να ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον υποψήφιο επίτροπο Βάλτης Δομπρόσκη σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ακρόαση ενώπιον των δύο επιτροπών μας δηλαδή έκον και έμπλο. Όπως γνωρίζετε, ο στόχος της ακρόασης ε, είναι να ασκήσει το δικαίωμά του το Κοινοβούλιο που απορρέει από τις συνθήκε να ψηφίσει για οποιοδήποτε ε, ομάδα επιτρέπων και ιδιαίτερα των μεμονωμένων επιτρόπων απαιτούνται ώστε να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους επιτρόπους επί τη βάση των γενικών τους ε, δυνατοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων, προσωπική τους ανεξαρτησία, ρεότητα, να, να, να αξιολογήσουμε τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, τις πολιτικές τους προτεραιότητες, τις ικανότητες τους να αναλάβουν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και τη ε, συμφωνία τους με τις νέες προτεραιότητες της νέας Επιτροπής. Να θυμίσω πριν την ακρόαση ότι ο υποψήφιος ε, Επίτροπος είχε γράψει είχε απαντήσει γραπτό σε ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Οι δε γραπτές του απαντήσει έχουν διανεμηθεί σε όλες τις γλώσσες του ευρωβουλευτέ και σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία ο υποψήφιος έχει υποβάλει και δήλωση συμφερόντων και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, είπε ότι δεν είχε καμία παρατήρηση όσον αφορά τη δήλωση συμφερόντων του υποψηφίου Επιτρόπου. Η διάρθρωση αυτής της ε, συζήτησης ε, θα γίνει ως ήθιστε. Καταρχήν ε, θα έχουμε μια πρώτη εισαγωγική δήλωση του υποψηφίου επιτρόπου, όχι πάνω από 15 λεπτά. 5 λεπτά θα έχει επίσης ο υποψήφιος επίτροπος για μια τελική δήλωση και Εν τω μεταξύ θα έχουμε τρία, τρίλεπτες ερωταπαντήσεις για τα μέλη. Ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Να θυμίσω επίσης ότι η αρχή των τριών λεπτών θα τηρηθεί αυστηρά, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η διερμηνία παρέχεται από 23 γλώσσες, ώστε όλοι οι ομιλητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και όπως είπα και σε άλλες ακροάσεις, θα σας ζητήσω να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να μπορείτε, ε, ώστε να, μπορείτε να μεταφραστείτε από τους διερμηνείς. Επί της ουσίας τώρα, τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο υποψήφιος επίτροπος Ντομπρόσκης είναι πάρα πολύ κέρια, δηλαδή να καθοδηγήσει τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, να κάνει τη διακυβέρνησή μας πιο συνεπή, αποτελεσματική, δημοκρατική και να αντιμετωπίσει την σημερινή οικονομική κρίση, επιτυχάνοντα σταθερότητα την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ εργάζεται σκληρά για να παρέχει τη συμβολή του Κοινοβουλίου σε μια γνήσια ατζέντα για την ΟΝΕ και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε την αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνηση Μαζί με εσά και του άλλου υπεύθυνου επιτρόπους θέλουμε να εντοπίσουμε τον καλύτερο τρόπο και της χρήσης ε, του κανόνα της ευελιξίας ώστε να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις και τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις να βελτιώσουμε την ε, οικονομική ε, τον συντονισμό και να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες διαφορές ανάμεσα στις αρμοδιότητες νομισματικής ε, πολιτικής και εκείνες ε, της οικονομικής πολιτικής και τέλος θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε και να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση μέσα στο πλαίσιο διακυβέρνησής μας. Αυτό το Κοινοβούλιο ζητά ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σύμφωνο. Και δίνω τώρα το λόγο στην Συμπροέδρο Μαρίζα ούσβολκ για να συνεχίσει αυτή την εισήγηση. Ορισμένα σχόλια εξ Επιτροπής ε, απασχόληση και αυτό το κάνω στα σουηδικά, ...στην μητρική μου γλώσσα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δυναμικό για να εγγυηθούμε την απασχόληση που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να ορίσει αυτούς τους όρους για την προστασία των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε μια κοινή αγορά που δεν θα πρέπει να μειώσει τις ε, καλές συνθήκες εργασίας ή να προβεί σε αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί αυτό θα μπορούσε να επαπειλήσει και τις ε, συλλογικές συμβάσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαχείριση της κρίσης στην αγορά εργασίας και θα πρέπει οι εταίροι να μπορούν να δράσουν αυτόνομα. Με την απόφαση Λαβάλ του δικαστηρίου βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για την ελεύθερη κυκλοφορία. Επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν είναι σοβαρές και χρησιμοποιούν τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιούνκερ, στην, στον ενακτήριο λόγο του μίλησε για την οδηγία περί αποσπασμένων εργαζομένων που θα πρέπει να επανεξεταστεί. Επίσης, αυτή η οδηγία θα πρέπει να αποτρέψει το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους μισθούς για την ίδια εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν υπεύθυνοι για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο. Ο κύριος Ντομπρόφσκης θα είναι υπεύθυνος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει υποσχεθεί πολλά. Οι εταίροι θα πρέπει να προωθήσουν και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις. Σε περίπτωση εκτροπών δεν μπορούμε να δεχτούμε μία άλλη οδό. Δεν μπορούν να ανταγωνίζονται τα κράτη-μέλη τα μεν τα δε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε τώρα το λόγο στον ε, κύριο Ντομπρόφσκης για 15 λεπτά το πολύ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σε εσάς, ε, τους ερετούς εκπροσώπους ε, των Ευρωπαίων. Το ότι ήμουν και εγώ δύο φορές ευρωβουλευτή. σημαίνει πως δεν χρειάζεται βεβαίως να μου υπενθυμίσετε την σημασία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν αναλάβω τελικά τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσω την πολιτική μας πρωτοβουλία και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των προτάσεών μας. Τα χαρτοφυλάκια μου είναι το ευρώ και ο κοινωνικός διάλογος. Θεωρώ λοιπόν πως τα καθήκοντά μου είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σταθερότητα, συντονισμός της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και βεβαίως στενότερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, γεννήθηκα και μεγάλωσα πίσω από το παραπέτασμα. Για 50 χρόνια η Λετωνία δεν μπορούσε να είναι μέρος της Ευρώπης δεν είχαμε βασικά δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Πριν από 25 χρόνια έπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα και έτσι άνοιξε ο δρόμος για ειρηνική δημοκρατική αλλαγή στην Ήπειρό μας. Η προοπτική για χώρες όπως η Λετωνία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατικής, οικονομικής και κοινωνικής μεταμόρφωσης. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω στη δύναμη του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Πιστεύω στις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής οικονομίας αγοράς και των ίσων ευκαιριών. Μόνο μαζί θα, μπορούμε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει γρήγορα, της παγκοσμιοποίησης, της γύρανσης και της κλιματικής αλλαγής. Είχα την τιμή να είμαι πρωθυπουργό Λετωνίας σε τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις από το Μάρτιο 2009 μέχρι και φέτος τον Ιανουάριο. Έλαβα καθήκοντα όταν η χώρα μου περνούσε την βαθύτερη οικονομική κρίση εντός της Ένωσης. Προτεραιότητα να αποκατασταθεί η ανάπτυξη και οι θέσει εργασία το συντομότερο δυνατόν. Ω αποτέλεσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, η Λετωνία βγήκε από την κρίση και έγινε μία από τις οικονομίες της Ευρώπης που αναπτύσσεται ταχύτερα. Υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, κυρίως ε, τα οικονομικά κίνητρα μέσω της ε, επιτάχυνσης της χρήσης των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων και δημιουργήσαμε ένα επιπλέον δίκτυ ε, κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης εκπληρώσαμε τα κριτήρια του Μάστριχτ και ενταχθήκαμε φέτος στο ευρώ. Αυτές οι διαδικασίες δεν θα ήταν δυνατόν να λάβουν χώρα χωρίς έναν διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους για τις ευαίσθητες πολιτικές και κοινωνικές αποφάσεις προετοιμαζόμενοι για την υιοθέτηση του ευρώ τη στιγμή που υπήρχε κρίση στην ευρωζώνη επιδείξαμε την εμπιστοσύνη μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το ευρώ τη στιγμή που άλλοι το αμφισβητούσαν. Στο παρελθόν ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος του ε, Λετωνικού Κοινοβουλίου, Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής οικονομολόγος της Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρώ πως η εμπειρία μου αυτή μου δίνει την απαραίτητη γνώση για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μπορώ να συνεισφέρω σε στην κοινωνική, οικονομική και νομισματική πολιτική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΟΝΕ και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα του ευρώ, να εργαστούμε προς μια σύγκληση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών με τις πολιτικές της αγοράς εργασίας. Εάν με εγκρίνεται λοιπόν στη θέση αυτή, θα εργαστώ σκληρά για να διαβασφαλίσω πως οι στόχοι της σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος και της μακροοικονομικής διακυβέρνησης θα συμβαστούν με την κοινωνική δικαιοσύνη και την συμπερίληψη όλων. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να αντιμετωπίσει τη χειρότερη κρίση στην ιστορία τη και να διαφυλάξει το ενιαίο τη νόμισμα. Αυτή τη στιγμή όμως ε, προβλέπεται πως τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτυχθεί με ένα 1,5% τα επόμενα 10 χρόνια όπως είπα. 1% λιγότερο δηλαδή από ό,τι στην προηγούμενη δεκαετία. Η κρίση εξακολουθεί λοιπόν να πλήττει τις κοινωνίες μας. Ε, στην Ευρωζώνη είναι πάνω από 11% η ανεργία, στους νέους είναι πάνω από 20% και 16% των Ευρωπαίων μεταξύ 15 και 29 δεν είναι ε, δεν έχουν ούτε δουλειά ούτε εκπαιδεύονται. Η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει μια ολόκληρη γενιά. Όλοι ξέρουμε πως ε, η κρίση αυτή δεν ήταν μια απλή μείωση των οικονομικών μεγεθών. Ε, οι αιτίες της ήταν αδυναμίες στις οικονομικές μας δομές. Γι' αυτό πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο με έναν πληθυσμό που γυράσκει με υψηλό επίπεδο χρέους και πολύ, χαμηλή, ε, πολύ χαμηλό πληθωρισμό η Ευρώπη να περάσει σε μια περίοδο χαμηλής ανάπτυξης ή ακόμα και στασιμότητας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους και να επανέλθουμε στο κατεύθυνση της αηφόρου ανάπτυξης. Οπότε χρειάζονται να αναλυθούν συγκεκριμένα και συντονισμένα μέτρα και από την πλευρά της ζήτηση και της προσφοράς και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει οι προτάσει της Κομισιόν να μεταφραστούν γρήγορα σε έργα. Αφετηρία θα είναι το επενδυτικό πακέτο 300 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων τα επόμενα τρία χρόνια και εδώ πέρα βέβαια συγκεκριτικό ρόλο θα παίξει ο αντιπρόεδρο για δουλειέ και ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται λοιπόν επενδύσει υψηλή ποιότητα για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για την υφιστάμενη χρηματοδότηση. Τα ευρωπαϊκά διαλευθερωτικά ταμεία πρέπει να επενδύονται σωστά και πρωτοβουλίε όπω η εγγύηση για την νεολαία πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Η κρίση κατέδειξε ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στον αρχικό προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου. Τα τελευταία χρόνια ελήφθησαν σοβαρά βήματα για την αντιμετώπιση τους. Η ε, δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση ενισχύθηκε. Επίσης ορίστηκε ένα πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης και υπάρχει μια εξάντε, ένας συντονισμός των εθνικών πολιτικών που ενισχύθηκαν υπό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίσης, ορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα ανάσχεσης τα τελευταία χρόνια. Η Τραπεζική Ένωση έχει καταλήξει και οι αδυναμίες των ισολογισμών των τραπεζών θα πρέπει να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να συνεχίσει η δανειοδότηση στην πραγματική οικονομία. Σήμερα είμαστε, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ πιο εύρωστη και μπορεί να οδηγήσει σε ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο που δεν προβαίνει σε κοινωνικούς αποκλεισμούς. Επίσης θα πρέπει να έχουμε έναν ευρύ κύκλο πολιτική συντονισμού το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έτσι ώστε να ορίσουμε συνεκτικές πολιτικές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το βαθμολόγιο απασχόλησης και κοινωνικών δικτών. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ευελιξία που ήδη υπάρχει στους κανόνες του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Θα πρέπει να έχουμε ίση μεταχείριση, να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών και διαχείριση κατά διαφανή τρόπο. Ο οικονομικός διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης ε, του χώρου του ευρώ μέσω του, του 2 και του 6 Εάν διοριστώ από το σώμα σας, θα αναλάβω όλα τα μέτρα έτσι ώστε να ενισχύσω αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την σταθερότητα και την αξιοπιστία μας μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών μας. Παράλληλα, θα πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή των συγκεκριμένων συστάσεων προς τα κράτη-μέλη θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα έτσι ώστε να έχουμε υψηλότερο επίπεδο η οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Θα πρέπει να μειώσουμε την ε, αδιαφάνεια στον τομέα των εισοδημάτων και την ανισότητα, καθώς και τη φτώχεια. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Αγαπητά μέλη, πιστεύω ότι η μελλοντική ανάπτυξη της ΟΝΕ αποτελεί έναν άμεσο αλλά και μεσοπρόθεσμο στόχο, όπως ορίστηκε από το προσχέδιο για μια πραγματική και αυθεντική ΟΝΕ. Έτσι θα μπορέσουμε να ε, προωθήσουμε την ΟΝΕ με βάση αυτά τα δεδομένα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στο μέτρο του δυνατού και να συμπεριλάβουμε στη συνεργασία αυτή και τα 28 κράτη-μέλη ο χώρος της Ευρωζώνης θα πρέπει να μείνει ανοιχτό σε νέα μέλη εάν πληρούνται τα κριτήρια του Μάστριχτ. Υπό αυτή την έννοια χαίρομαι διότι η Λιθουανία θα γίνει το 19ο μέλος της Ευρωζώνης στους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό αφορά βέβαια και τη χρήση της κοινοτικής μεθόδου. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις διάφορες επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την ενδεχόμενη αλλαγή των συνθήκων. Αγαπητά μέλη, και αν διοριστώ αντιπρόεδρος, η εντολή μου θα αφορά μία εργασία για την επανεξισορρόπηση των όρων σταθερότητας μέσα στα πλαίσια των χωρών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ε, Δέχουμε τη δέσμευση του Προέδρου Γιούνκερ μέσα στα πλαίσια της ε, δημοσιονομικής συνεργασίας και αποτίμησης. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί κράτη-μέλη να προστρέξουν σε τέτοια προγράμματα πλέον τη στιγμή που ορίστηκε η Τρόικα και διορίστηκε για να διαχειριστεί μια κατάσταση οικονομικής καταστροφής θα πρέπει στη συνέχεια να, να, να αντικατασταθεί από νέα νόμιμα δημοκρατικά μέσα και διαφρόσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και να ασχοληθούμε και με τις δύο πλευρές του νομίσματος, δηλαδή το οικονομικό σκέλος και το κοινωνικό. Διαμέσω της ιστορίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κοινωνικού διαλόγου Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ε, ανταλλαγές απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους επί της ουσίας. Ο κοινωνικός διάλογος είναι απόλυτα αναγκαίος έτσι ώστε οι μεταρρυθμίσεις να καταστούν δυνατές και βιώσιμες. Είναι ένα απαράβατος όρος για την ευημερία της ΟΝΕ. Θα συνεργαστώ με τους Επιτρόπους Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και κινητικότητας ε, της αγοράς για να ενισχύσουμε αυτά τα μέτρα και σε εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος ε, του Αντιπροέδρου για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο αποτελεί απάβγασμα του στόχου του Προέδρου για την ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άμεση συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας για να προωθήσω την οικονομική και, κοινωνικό, και κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης και ξεκινάμε αμέσως με το πρώτο γύρο των ομιλητών με τον κύριο Μπάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντομπρόφσκης. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ πέρα με την πολιτική σας στην χώρα σας νομίζω είχατε σοβαρές επιτυχίες και τελικά μπόρεσε η χώρα σας να μπει στην ΟΝΕ. Και μάλιστα μπόρεσα να τα διαπιστώσω όλα αυτά από πρώτο χέρι γιατί ήμουν ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξη της Λετωνίας στο ευρώ. Καταφέρατε σε λίγα χρόνια να περάσετε την Λετωνία από χώρα προβληματική ε, σε μια χώρα με ελάχιστο έλλειμμα του προϋπολογισμού και σαφώς καλύτερα στοιχεία γνωρίζουμε και ελπίζουμε πως θα το συνεχίσετε αυτό στο μέλλον. Οπότε το ερώτημά μου είναι ποια είναι για σας η, επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική μεταρρυθμίσεων και τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε και υγιείς προϋπολογισμούς και περισσότερη ανταγωνιστικότητα και ποιο ρόλο βλέπετε εδώ πέρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Κύριε Μπάλτς. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την περτέρω εξέλιξη της Ένωσης και της ΟΝΕ, νομίζω πως σταδιακά περνάμε από τη φάση της δημοσιονομικής προσαρμογής που έγινε όχι παντού, αλλά σε γενικές γραμμές έχει γίνει παντού, στη φάση στην οποία πρέπει να έχουμε μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε κάποιους παράγοντες, κυρίως προς τρεις κατευθύνσεις. Το ένα είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και των κρατών μελών, να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά ειδικά σε τομείς όπως υπηρεσίες, ενέργεια, ψηφιακή ενιαία αγορά. Να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη γνώση, γιατί η έρευνα και η καινοτομία είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου οι άλλες προηγουμένες οικονομίες ξοδεύουν περισσότερα, να μειωθεί το διοικητικό βάρος και η γραφειοκρατία, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. χρειάζονται επενδύσεις και το ανέφερα πως μία από τις βασικές προτεραιότητες τη Νέας επιτροπή είναι να προετοιμάσει ένα πρόγραμμα 300 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων τα επόμενα τρία χρόνια και πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και βεβαίως η πλευρά της ζήτησης στην οικονομία, γιατί αυτά τα πράγματα συνδέονται. Η ε, οικονομική σταθερότητα, επενδύσεις και ζήτηση. Και με τις τρεις αυτές πτυχές θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ελίζα Φερέιρα τώρα, συντονίστρια των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Όπως ξέρετε η Ευρωζώνη και κυρίως τα νοτιότερα μέλη της ε, αντιμετωπίζουν μια κρίση άνευ που δεν μπορούν να την αντιμετωπίζουν αυτή τη φάση της ύφεση και της ψηλής ανεργίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ε, τυφλής πολιτικής λιτότητας ε, του τύπου που εσείς ως Πρωθυπουργό της Λετωνίας εφαρμόσατε στη δική σας χώρα πολύ πιο, σε πολύ πιο βέβαια πλαίσιο από ό,τι το σημερινό. Ε, πώς μπορείτε να μας πείσετε ότι αλλάξατε και ότι σήμερα είστε γνήσιος και δεσμευμένος ερμηνευτής της αλλαγής της στην οικονομική ατζέντα, όπως αυτή την υποσχέθηκε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Τι είδους συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε έτοιμος να αναλάβετε για το μέλλον, που μας δείχνουν ότι αν κυρωθείτε δεν θα επιστρέψετε στην στάση λιτότητας και πώς ερμηνεύετε το καταμερισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε εσά και τον υποψήφιο επίτροπο ε, Μοσκοβισή. Ευχαριστώ κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας που ήταν οι τρεις και θα είμαι πολύ σύντομος για να μπορέσω να απαντήσω και στις τρεις πτυχές. Ε, Όσον αφορά τις γενικές κατευθύνσεις της εργασίας της Κομισιόν, καθώς επίσης και τις δεσμεύσεις, προσπάθησα να τις τονίσω να, στις μου παρατηρήσεις και συνυπογράφω απόλυτα την προσέγγιση του υποψηφίου προέδρου, του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γιούγκερ ότι δηλαδή ενώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε οικονομικές και νομισματικές πολιτικές θα πρέπει ταυτόχρονα να αναλάβουμε και τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Είμαι απόλυτα έτοιμος να συνεργαστώ και να εργαστώ σε αυτές τις γραμμές και ακριβώς θεωρώ πως αυτό είναι το καθήκον μου και στην εκτέλεση του καθήκοντός μου ε, σκοπεύω να συνεργαστώ στενά τόσο με τον Επίτροπο Μοσκοβίτσι όσο και με τον υποψήφιο, ε, ε, την υποψήφια Επίτροπο Τάισεν ώστε να συνδυάσουμε τα οικονομικά με τα κοινωνικά θέματα. Όσον αφορά τον τρόπο συνεργασίας, ξέρουμε ότι αυτή είναι μια νέα πρόταση του, του Προέδρου Γιούγκερ να υπάρξει δηλαδή ένα συντονιστικός ρόλος, αλλά είναι σαφές πως εμείς αυτό το βλέπουμε ως συλλογική εργασία. Δεν το βλέπουμε ε, ότι υπάρχει κάποια ιεραρχία. Το έχουμε συζητήσει και με τον υποψήφιο επίτροπο Μοσχοβίτσι και νομίζω πως μπορούμε κάλλιστα να βρούμε τρόπο συνεργασίας. Δεν σημαίνει αυτό με κανένα τρόπο ότι υποβαθμίζουμε το έργο ενός ή άλλου επιτρόπου, ενώ ο Πρόεδρος θα συντονίζει τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές και θα μεριμνεί ώστε να συμβαδίζουν. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Κέιτ Σουίμπορν, που είναι συντονίστρια του ECR στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ και καλώς ορίσατε υποψήφια τον Πρόσχη. Το βιογραφικό σας λέει ότι είστε, έχετε πάρα πολλά προσόντα και ότι αντιστοιχείτε στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως Αντιπρόεδρος για το Ευρώ και το Κοινωνικό Διάλογο θα έχετε πολύ ευρία εντολή και γι' αυτό και η ερώτησή μου είναι το ίδιο ευρία. Ως εκπρόσωπος της Ένωσης στα διάφορα διεθνή φόρα βήματα όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι θα πείτε στους διεθνούς ομολόγους ε, ότι είναι οι ε, προτεραιότητες σε μέσο και βράχη πρόθεσμα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ευχαριστώ πολύ. όσον αφορά τις εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνή βήματα όπως ε, το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Σταθερότητας ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία έχει θέσει η το διεθνες ομισματικο ταμειο υπαρχουν διαφορα ζητηματα Ένωση ως προτεραιότητες όσον αφορά την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχουμε θεσπίσει προτεραιότητες. Πρόκειται για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής. Ε, αυτό το τονίζουμε πολύ στους διεθνείς μας εταίρους. Γνωρίζουμε ότι γίνονται επίσης συζητήσεις για την μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πιστεύω και ότι από την πλευρά της Ένωσης χρειάζεται να συντονίσουμε ε, έντονα τις θέσεις των διαφόρων κρατών μελών που αντιπροσωπεύονται στον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί τα κράτη τη Ένωση είναι αυτά που εδράζουν στο Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και που συμμετέχουν σε συνεδριάσει αυτού. Τώρα, όσον αφορά το FSB, το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει εκεί να γίνει είναι να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία περί οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι διάφορες χώρες και διάφορες περιφέρειες συχνά ακολουθούν προσεγγίσεις ή συντάσσουν νομοθεσίες που έχουν εξωεδαφικές εφαρμογές ή επιρροές. Ε, δηλαδή εκτός της επικράτειάς τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπειες και επικάλυψη. Αυτό που θέλουμε να, να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν σαφείς αρχές για το πώς, ε, ε, πώς εφαρμόζεται η οικονομική διακυβέρνηση έτσι ώστε οι, οι διάφορες χώρες και οι διάφορες περιφέρειες να μην προσπαθούν να κάνουν η καθεμία το δικό της με τρόπους αντικρουόμενους μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Τώρα ε, η Άλντι Σιλβί Γκουλάρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ναι, βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που αναφέρατε ρητά τον ε, στόχο της καταπολέμησης της στόχιας. Ε, αυτό είναι πολύ ευτυχές, γιατί δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα πείτε μου ακριβώς πώς θα συνεργαστείτε με το Πιέρ Μοσκοβισή. Εγώ δεν κατάλαβα μέχρι τώρα. Πρέπει να λάβετε κοινά αποφάσεις για τα θέματα εφαρμογής κανόνων αλλά προέρχεστε από δύο τελείω διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα. σω να μου πείτε, ότι, όπως μας είπε και εκείνο, ότι θα δουλέψετε ομαδικά και εμεί μα αρέσουν οι αγαπημένοι επίτροποι, αλλά εν πάση περιπτώσει συγκεκριμένα τι θα κάνετε. Θα επιτρέψετε σε κάποιες χώρε που δεν τηρούν ε, τους κανόνες ε, να λάβουν υπόψη ας πούμε, τις, δαπα... τις επενδυτικές δαπάνες και έπειτα για τα όσα γίνονται εκτός Ένωσης. Ποιος θα αντιπροσωπεύει την Ευρωζώνη στα διεθνή φόρα, η επιστολή του κύριου Γιούγκερ μας μίλησε για δεσμεύσεις πραγματικέ και ρεαλιστικές. Εσείς μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ κυρία Γκουλάρ για την ερώτηση αυτή. Και πάλι δεν ήταν μία, ήταν ε, διάφορες ερωτήσεις μαζί. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον υποψήφιο επίτροπο Μοσχοβησή. Όπως έχω ήδη δηλώσει και όπως και ο ίδιος δήλωσε κατά τη διάρκεια της δικής του ακρόσης επανελειμμένα, είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να, εργαστούμε, να συνεργαστούμε στενά, σε πνεύμα ε, αγαστής συνεργασίας και ούτω ή άλλω οι επίτροποι προέρχονται από διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Και ωστόσο, η, αλλω οι επιτροποι προερχονται απο διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. και ωστοσο η ομαδα η, η Κομισιόν πρέπει να εργαστεί ω ομάδα και άρα πρέπει να αφήσει στην άκρη τι διαφορέ του καθένα και να εργαστεί για την επίτευξη ενό κοινού ε, σκοπού. Και αυτό θα κάνουμε και με τον ε, κύριο Μοσκοβίση. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχουμε συμφωνήσει. Τώρα, για την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης. Όπως είπατε σωστά, ο πρόεδρος Γιούνκερ θα πρέπει να βρει κάποιες ρεαλιστικές ρυθμίσεις όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση οι υπεύθυνοι επίτροποι θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους συμπεριλαμβανομένου του έργου της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ένωσης. Ήδη δηλαδή έχουμε συζητήσει αυτή την επιτυχή εξωτερικής εκπροσώπησης με τον υποψήφιο επίτροπο Μοσκοβισή. Έχουμε συμφωνήσει επί των γενικών αρχών και αυτή τη στιγμή τα επιτελεία μας συνεργάζονται ώστε να ε, να καταλήξουν μάλλον στις πρακτικές ρυθμίσεις που θα υποβληθούν στις πρώτες και όλες τις εβδομάδες της εντολής μας, όπως μας ζήτησε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Σε ευχαριστώ για την Γκουή Μιγγέλ Βιέγκας. Ε, Απλή ερώτηση. Βλέποντας την ιστορία του ευρώ, τα τελευταία 14 χρόνια βλέπουμε ότι από τα 28 κράτη-μέλη τα 23 δεν τήρησαν τους ε, κανόνες για το δημόσιο χρέος. Επίσης το βαθμολόγιο δείχνει ότι κανένα, καμία χώρα δεν πληρεί τις ε, μακροοικονομικές ε, προϋποθέσεις και η χώρες εκτός Ευρωζώνης αναπτύσσονται περισσότερο και έχουν χαμηλότερο χρέος από τις χώρες της Ευρωζώνης. Μπορούμε να κάνουμε και διεθνείς συγκρίσεις και να δούμε ότι άλλες περιοχές της παγκόσμιας σχακέρας έχουν ένα ρυθμό ανάπτυξης τρεις φορές υψηλότερο. Άρα πώς μπορούμε να φτάνουμε σε μια κατάσταση εκτός νομιμότητας και να ορίσουμε νέους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης. Κύριε καταρχήν σε σχέση με τις ε, χώρες ε, που βρίσκονται σε μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τις, 23 ε, χώρες έχουν, ε, ε, έχει μειωθεί ο αριθμός. Δηλαδή οι χώρες είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι 3-4 χρόνια πριν. Αλλά πολύ σωστά αναφέρατε ότι σε σχέση με άλλες προηγμένες οικονομίες, οι άλλες οικονομίες ανακάμπτουν με ταχύτερους ρυθμούς. Γι' αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε τις πολιτικές μας και να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι για κάτι τέτοιο. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα ως προς τις επενδύσεις μεταξύ το 2009 του 8 και 9 οι επενδύσεις της ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσαν κατά 19%. Είχαμε ίδια σημεία εκκίνηση. Το 2013 οι επενδύσεις της ΕΠΑ αυξήθηκαν κατά 34% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 3% αντιστοίχως σε σχέση με το 9%. Εάν θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε σε μια οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις και τη ζήτηση. Η χρηματοοικονομική σταθερότητα αποτελεί πρόκριμα για την ανάπτυξη, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και γι' αυτό η νέα Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση των χωρών εκτός Ευρωζώνης, γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι μακροοικονομικές διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος ισχύουν σε, για όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο της μακρονομικής διακυβέρνησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός και εκτός Ευρωζώνης. Γκίγκολτ. Κύριε συνάδελφε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είπατε τόσο πολλά πράγματα για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Το τελευταία χρόνια είδαμε ε, μείωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Τρόικας ε, αλλά και με βάση τα όσα έκανε και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για να, για να προετοιμάσει τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Δεν είναι διαφανή αυτά τα θεσμικά όργανα και δεν είναι υπόλογα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε στην Τρόικα, θα ήθελα όμως να γνωρίζω συγκεκριμένα τι μέτρα θα λάβετε για να δημιουργήσετε διαφάνεια σε όλα τα θεσμικά όργανα και να υπάρχει και δημοκρατική ευθύνη και λογοδοσία. Και θα ήθελα το δεύτερο ερώτημα να μου πείτε εάν είστε διατεθειμένος να προετοιμάσετε μια διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπολείπων τμήματων της λεγόμενης οικονομικής διακυβέρνησης για να υπάρξει κάποια ενίσχυση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Πρώτα απ' όλα για τη δημοκρατική νομοποίηση της Τρόικας. Ανέφερα ήδη το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει όταν δηλαδή ε, δίνονται κάποιες ε, σύμβουλες στις χώρες ε, του προγράμματος να μην γίνεται μόνο οικονομική αξιολόγηση αντικτύπου αλλά αξιολόγηση αντικτύπου και των κοινωνικών πτυχών και των πτυχών της απασχόλησης για να δούμε πώς επηρεάζει όλους τους δείκτες αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μετά για το επόμενο σαφώς πρέπει να υπάρχει περισσότερη λογοδοσία και οπωσδήποτε και αυτό είμαι διατηθειμένος να το συζητήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με άλλους εμπλεκόμενους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να είμαστε να έχουμε περισσότερη λογοδοσία. Είναι σαφής δέσμευση αυτή του Πρόεδρου Γιούνκερ και συμφωνώ πλήρως για τον ρόλο του Eurogroup στην ε, λήψη αποφάσεων. Οπωσδήποτε για την Κομισιόν είναι δύσκολο να συζητήσουμε τα εσωτερικά άλλων ε, θεσμικών οργάνων. Γιατί τώρα μιλάμε για το πώς λειτουργεί το Συμβούλιο. Αλλά ως ε, γενικό κανόνα θα έλεγα πως ε, σαφώς πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε στόχο να αναπτυχθούν και 28 χώρες. Άρα ο ρόλος του Eurogroup πρέπει να σχετίζεται με το ευρώ. Ενώ ευρύτερα μακροοικονομικά ζητήματα, ζητήματα εσωτερικής αγοράς πρέπει να τα αντιμετωπίζει το ΕΚΟΦΗΝ. Για την τρίτη ερώτηση θα σας απαντήσω κάποια άλλη στιγμή για τη διοργανική συμφωνία. Τελείωσε ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ. Πάτρικ Οφλίν για το EFTD. Κύριε Ντομπρόφσκης, στις γραπτές σας απαντήσεις μιλάτε για την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Λέτε πως η Οικονομική και Ένωση πρέπει να γίνει πιο συνεκτική, να έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση στο σύνολο της Ένωσης αναφέρεται κάποιες απαιτήσει για τις εθνικές κυβερνήσεις για να λειτουργεί καλύτερα το ευρώ. Και σαφώς εδώ πέρα συμφωνεί με αυτά ο κύριος Ντράγκη, αλλά μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες πώς θα επιβάλλετε αυτή την σύγκληση χωρίς να υπονομεύσετε την εθνική δημοκρατία αν περιορίζετε τα ζητήματα που θα κρίνονται στις εκλογές και εναλλακτικά γιατί η α, αντίστοιχη πορεία είναι αδιανόητη για εσάς, δηλαδή να έχουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ευρώ και να επανέλθουν οι κεντρικές τράπεζες και τα εθνικά νομίσματα. Και έτσι όπως πάει το ευρώ μέχρι στιγμής, αναρωτιέστε ποτέ μήπως η εναλλακτική την οποία ανέπτυξα θα ήταν καλύτερη και από πλευράς δημοκρατίας και από πλευράς οικονομικής απόδοσης πολλών χωρών. Εντάξει, τελείωσε ο χρόνος σας λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Για την πρώτη σας ερώτηση της ε, σύγκλησης της πολιτικής ε, και της ε, διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Αυτό γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπου παρουσιάζουμε τις βασικές κατευθύνσεις των επόμενων 18 μηνών και με βάση αυτό προετοιμάζουμε τις ε, συστάσεις μας αναχώρα. Έτσι, βασικά, λειτουργεί η διακυβέρνηση αυτή. Βεβαίως είναι κάτι το περίπλοκο που περιλαμβάνει πολλές άλλες πτυχές. Μετά, σαφώς δεν συμφωνώ με την απόψή σας ε, για τα ωφέλη της διάλυσης ε, της ε, Ευρωζώνης. Εγώ θεωρώ πως το ευρώ ήταν τεράστια επιτυχία παρά την κρίση και πράγματι ε, η Λετωνία είχε τεράστια οικονομική κρίση το 2008-2009 ε, χωρίς το ευρώ και άλλες χώρες εκτός της Ευρωζώνης το ίδιο. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι το ευρώ. Αν δείτε το ευρώ ως νόμισμα, μια χαρά τα πάει. Ε, η ισοτιμία του είναι πιο κοντά στο ιστορικό ύψιλο, ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα παραμένει σταθερό, ε, ένα τέταρτο των παγκοσμίων αποθεμάτων είναι σε ευρώ, οπότε σαφώς όταν μιλάμε με οικονομικά, για οικονομικά προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν πρέπει πάντα να τα ρίχνουμε στο ευρώ. Μάλιστα για τους μη εγγεγραμμένους ο Μπερνάρ Μονό. Δώδεκα χρόνια μετά από την ε, ΟΝΕ βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές ε, και μιλάμε για μια ευρωζώνη που είναι η ζώνη του απόλυτου μηδέν γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει μια τέτοια ευρωζώνη. Εδώ και τέσσερα χρόνια θα πρέπει να εξεύρουμε σχέδια διάσωσης, ακόμα και για τη Γαλλία που είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρώπης, μιλάμε για ένα χρέος 520 δις ευρώ. Άρα δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι δυστυχώς το έλλειμμά μας γίνεται ολοένα και πιο ε, εξωφρενικό εσείς. Δεν δέχεστε να, να γίνεται υποτίμηση, αλλά στη δική σας χώρα έγινε ε, μία μείωση μισθών κατά 20% για να ανταποκριθείτε. Μετά το 2008, την Πανελλονιωθρία τη Μεγάλη ή στην Κύπρο το 2013, πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε γιατί ακόμα και η αγορά του χρέους από την ΕΚΤ δεν επαρκεί. πώς θα προωθήσετε λοιπόν τον κοινωνικό διάλογο προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως είπε, ήδη σας είπα στη εισήγησή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη γνώρισαν τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία τους. Αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη αντιμετώπισαν αυτή την κρίση και βγήκαν πιο δυνατές μετά την κρίση αυτή. Και οι αρχικές αδυναμίες αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με την αρχικά προγραμματισμένη ΟΝΕ. Βλέπουμε επίσης ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν έγιναν αποδοτικές μέσα στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής σταθερότητας. Φέτος επανερχόμαστε στην οικονομική σταθερότητα και του χρόνου για πρώτη φορά μετά την κρίση όλα τα κράτη-μέλη θα ε, έχουν θετική ανάπτυξη. Βεβαίως υπάρχουν δύσκολα θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν στην Ευρωζώνη. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πιο δυνατοί αν αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα από κοινού ή αν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ξεχωριστά διαλύοντας την Ευρωζώνη. Γι' αυτό και δεν δέχομαι τη δική ε, το δικό σας σκεπτικό για την κατεύθυνση που πρέπει να ε, ακολουθήσουμε. Δεύτερος γύρος, εξ ονόματος των Επίτροπων, ο David Κάζα, λόγο από το ΕΛΚ. Κύριε ε, υποψήφιε επίτροπε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στρέφεστε προς τις ευρωπαϊκές αξίες και ξέρω ότι είναι εύκολη συνεργασία μαζί σας. Όμως είπατε ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ίσως αντικαταστήσει την Τρόικα με μια νέα διάρθρωση, η οποία θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν κοινωνικό πρόσωπο και θα προωθήσει το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αξιολογήσεις κοινωνικού περιεχομένου για να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε αυτή την, την κοινωνική αποτίμηση, η συνολική αξιολόγηση στην οποία αναφερθήκατε. Τον Ευχαριστώ κύριε Κάσα. Μου υποβάλατε δύο ερωτήσεις ως προς την πρώτη. Για τις διάφορες διευθετήσεις επί του συστήματος της Τρόικας και κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί στην κοινοτική μεθοδολογία ή πλαίσιο, αυτό είναι κάτι που γίνεται δεκτό από την Επιτροπή και θέλουμε να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να γίνουν μακροοικονομικές οικονομικές διευθετήσεις και να ενταχθούν στην κοινοτική μέθοδο. Αλλά γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Και αν και πρέπει να αντιδράσουμε και χρειάστηκε να ανταποκριθούμε άμεσα με την έναρξη της κρίσης, τότε δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μία αλλαγή των συνθήκων, γιατί λόγω κρίσης έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Γι' αυτό πολλά επιλήθηκαν διακυβερνητικά. Όμως θα ενταχθεί το σύστημα της ε, Τρόικας στην κοινοτική μέθοδο ως προς την ε, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην οικονομική διακυβέρνηση τις τελευταίες ε, εβδομάδες. Ήρθα σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους για να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή ιδεών και θεωρώ ότι θα πρέπει να τους φέρουμε πιο κοντά στο ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο. Και εδώ μιλώ για, το ευρωπαϊκό επίπεδο που γίνονται συζητήσεις με τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Και κατά τη μελέτη ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα αυτό. Και σε εθνικό επίπεδο με βάση τις συστάσεις προς την κάθε χώρα ξεχωριστά. Αυτή θα είναι η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο Πέτερ Ζήμων από τους σοσιαλιστές. Ναι, κύριε Ντομπρόφσκης, ε, από ό,τι φαίνεται θα αναλάβετε, προτείνεστε μάλλον για αντιπρόεδρος για το ευρώ και την κοινωνική συνοχή, αλλά βεβαίως ε, βλέπουμε πως ε, πάρα πολλές χώρες είτε υπό την Τρόικα, είτε η δική σας η χώρα χωρίς την Τρόικα έκανα κάποιες μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν σε καταστροφικές συνέπειες. Θεωρώ λοιπόν πως για την ομάδα μου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η απάντηση της εξής ερώτησης. Συμφωνείτε πως τα προγράμματα λιτότητας ε, που επιβλήθηκαν από την Τρόικα είναι βασικές ουσίες για τις τραγικές κοινωνικές συνθήκες της χώρες αυτές. Δεδομένης της σημασίας της ερώτησης αυτής για την ε, ομάδα μου σας παρακαλώ να είστε σαφείς και να απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι και μετά πείτε μου τι ρόλο έπαιξε και θα παίξει αυτή η αξιολόγηση για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των προγραμμάτων αυτών. Μάλιστα. Βεβαίως είναι ε, ένα ζήτημα περίπλοκο. Οπότε όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική κρίση δεν ε, τίθεται ζήτημα για το ότι πράγματι η κρίση δημιούργησε κοινωνικά προβλήματα και αύξησε την ανεργία ουσιαστικά. Υπάρχει, νομίζω όμως, ε, περιθώριο συζήτησης για τις αιτίε και τις συνέπειες. Γιατί γνωρίζετε πως η πολιτική λιτότητας, κατά μία έννοια, ήταν συνέπεια της κρίσης. Δεν ήταν ότι οι χώρες πήγαιναν μια χαρά και είχαν πρόσβαση στις αγορές και ξαφνικά αποφάσισαν να κάνουν κάποια δημοσιονομική προσαρμογή. Γεγονός ήταν πως οι χώρες είχαν σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες και η χώρα μου, η Λετωνία, και είχαν βρεθεί εκτός αγορών και έπρεπε να αντιδράσουν ε, με τρόπο γρήγορο, άμεσο δηλαδή. Βεβαίω μπορεί κανείς μετά πάντα να εξετάσει το εάν όλες οι αποφάσεις που ελήθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και στη Λετωνία ήταν οι σωστές. Και βεβαίως εκ των υστέρων πράγματι μπορούμε να βρούμε αρκετά λάθη. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα λάθη για να αποφύγουμε αυτό το σενάριο που ανέφερα ότι αντιμετωπίζουμε πολύ χαμηλή ανάπτυξη ή και στασιμότητα και να το μετατρέψουμε σε ένα σενάριο αηφόρου ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ, Ρόμπερτ Ζέλε, για το ECR. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Τσίλε. Λειτουργεί. Ε, αλλάξτε θέση αν δεν λειτουργεί εκεί το μικρόφωνο σας. Κύριε Ντομπρόφσκης, ε, αναφέρατε βεβαίως το ότι ήσασταν στην κυβέρνηση κατά την διάρκεια των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στην χώρα σας. Εγώ όμως θα ήθελα να αφαιρθώ στον κοινωνικό διάλογο. Συχνά μιλάμε για το κοινωνικό ντάμπινγκ για ένα κομμάτι της, ε, του ανοίγματο της αγοράς υπηρεσιών. Βλέπουμε πως ε, συχνά δεν πληρώνεται ο ίδιος μισθός για την ίδια εργασία σε διάφορες χώρες. Θεωρείτε λοιπόν πως υπάρχει κάποια δυνατότητα δημιουργίας ενιαίας αγοράς της υπηρεσίας ή βλέπετε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και το θέμα του κοινωνικού dumping. Πρώτα απ' όλα, αν μιλάμε για τρόπους ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου νομίζω πως ε, όλες οι προτεραιότητες ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μας φανούν χρήσιμες. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τα ζητήματα, τα εγγενή στην ε, μακροοικονομική τη λεγόμενη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης για το ερώτημά σας συγκεκριμένα όσον αφορά την εσωτερική αγορά υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα που ανέπτυξα στην αρχή μου δήλωση. Μιλάμε για ενέργεια, υπηρεσίες, ψηφιακή ενιαία αγορά. Όλα αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να το δει αυτό το ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά την ε, οδηγία περί απόσπασης ε, εργαζομένων. Πράγματι συχνά τίθεται το ζήτημα του κοινωνικού dumping και σκοπεύουμε να αναθεωρήσουμε την οδηγία για να μπορούμε να δούμε πού ακριβώς δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, πώς ερμηνεύονται οι κανόνες ε, περί βασικού μισθού. Υπάρχουν ζητήματα που μπορούμε να δούμε. Μια, τρόπο είναι μια νέα οδηγία που θα αφορά ακριβώς την εφαρμογή της απόσπασης εργαζομένων. Και βεβαίως μετά, αν περάσει, θα γίνει νόμος και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ. Από την Αλντε, Γιώχαν Χάιζεν. Κύριε υποψήφιε Επίτροπε, ο πρόεδρος ε, της ΕΚ, ο κύριος Ντράγκη, στις 22 Σεπτεμβρίου στην ΕΚΟΝ, είπε ότι καμία νομισματική πολιτική δεν έχει νόημα χωρίς να υπάρχει και η αντίστοιχη δημοσιονομική πολιτική. Ε, δέχεστε αυτή τη δήλωση και τι πιστεύετε στην περίπτωση της ποσοτικής ελάφρυνσης. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, στη γραπτή σας απάντηση είπατε ότι θέλετε να αυξηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε εθνικό επίπεδο, αλλά όταν συζητήσαμε με άλλα κοινοβούλια ε, για το θέμα του εξαμήνου, πολλές χώρες δεν ήταν καν παρούσες, για παράδειγμα η Ελλάδα και η Γερμανία. Άρα, ποια είναι τα σχέδιά σας σε σχέση με την ανάπτυξη αυτού του καθεστώτος σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. σε σχέση με το ρόλο της ΕΚΤ και τι μπορεί να κάνει μία νομισματική πολιτική και μία καθαρά δημοσιονομική. Βεβαίως χρειαζόμαστε σαφείς πολιτικές και νομισματικής υφής και δημοσιονομικής. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο τη μία ή την άλλη. Είναι ένα θέμα που αφορά ε, τα διάφορα ε, σκέλη του μηχανισμού λύσης αποφάσεων. Ως προς την ποσοτική ελάφρυνση, η ΕΚΤ αυτή τη στιγμή προβάλλει μία νομισματική πολιτική με επιτόκια πάρα πολύ χαμηλά ιστορικά πιο χαμηλά, σε ιστορικά πιο χαμηλά επίπεδα και σε σχέση με την ε, ποσοτική ελάφρυνση, εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, περίπτωση ευρωομολόγων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ή συνθήκες που δεν πληρούνται και η ΕΚΤ ζήτησε την αγορά συγκεκριμένων ομολογιών για να μπορέσει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τους ισολογισμούς τους. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να γίνει μια εισβάθος μελέτη πριν από συγκεκριμένες συστάσεις προς ε, τα κράτη-μέλη, μεμονωμένα δηλαδή. Παλώμα Λόπες, Γκουε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκης, η χώρα σας είναι η πιο άνηση. Βλέπουμε ότι λόγω της απασχόλησης, της χαμηλής απασχόλησης, πολλοί οδηγήθηκαν στη μετανάστευση εξαιτίας της ε, πολιτικής σας λιτότητας. Μιλάτε για έλεγχο της ευρωπαϊκής οικονομίας, όμως τα μέτρα σας δεν θα είναι αποδοτικά τη στιγμή που προβάλλεται μια πολιτική οικονομικής λιτότητας πώς ε, θα προωθήσετε τον κοινωνικό διάλογο που σταμάτησε μονομερός η τρέχουσα επιτροπή. Πρέπει να προωθήσουμε καλύτερους μισθούς και αξιοπρεπή εργασία. Επίσης, η, κοινότητα χρειάζεται επενδύσεις ε, πάνω από 300 δις. Επίσης, ε, πώς το Six Pack θα λάβει υπόψη την κοινωνική συνοχή της Ευρωζώνης. Και πάλι να σας πω ότι πρόκειται για τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν για τις προτεραιότητες. Αυτό που η νέα Επιτροπή θεωρεί προτεραιότητα είναι ακριβώς να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενώ παρέχει ε, παραδοσιακές επενδύσεις. Αυτό δεν θα το ε, δεν θα ήθελα να, το, ε, να πω ότι τα 400 δισεκατομμύρια αυτά είναι ανακύκλωση παλιών χρημάτων. Όχι, δεν είναι αυτή η πρόθεση της Κομισιόν. Είναι, η πρόθεσή μας είναι να έχουμε μια φιλόδοξη πρόταση που θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης. δημοσιονομικές προσαρμογές έχουν γίνει. Πρέπει να εστιάσουμε στην πλευρά της ζήτησης και με την αύξηση των μισθών. Αν δεν θέλουμε να χάσουμε την ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα είναι σημαντική. Θα πρέπει να αλλάξουμε τη φορολόγηση, να μετακινήσουμε τη φορολόγηση από την εργασία, ιδιαίτερα την χαμηλόμιστη εργασία, στο κεφάλαιο στην ιδιοκτησία και έτσι να, μπορέσουμε, να μπορέσουν να δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης. Όσον αφορά τώρα το διπλό και το εξαπλό πακέτο, αναφέρω μια από τις επιλογές για το πώς θα εξασφαλίσουμε περισσότερη κοινωνική σύγκληση, δηλαδή θα λάβουμε υπόψη τους δείκτες, τους κοινωνικούς και τους δείκτες απασχόλησης που εντάζονται στην νομοθεσία και που αυτή τη στιγμή χρησιμεύουν ως βοηθητικοί δείκτες. Σας ευχαριστώ. Thank you. Η κυρία Τατιάνα Ζδάνοκα των Πρασίνων είναι η επόμενη ε, ομιλήτρια. Εδώ βρίσκομαι. Τρεις συναδελφοί τουλάχιστον ρώτησαν για την Τρόικα. και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να, τον, ε, να την μετατρέψει ο πρόεδρος Γιούνκερ. Τρεις ε, λοιπόν ρώτησαν. Εσείς έχετε εμπειρία σε αυτό το τομέα. Γιατί η κυβέρνηση της οποίας εσείς ηγηθήκατε υιοθέτησε δραστικές ε, περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στους όρους που του εισετέθησαν. Ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τα πόσο ήταν δική τους επιθυμία ή δική σας απόφαση να τα βγάλετε όλα πέρα με στο πλάτη των ε, ε, πολιτών. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, Δύο ερωτήσεις όσον αφορά το ρόλο της Τρόικα. Το πρώτο βήμα στο οποίο θα πρέπει να προβούμε, πρόθεσμα, είναι ότι οποιαδήποτε πολιτική οθετηθεί όχι μόνο θα πρέπει να ταιριάζει με τη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό αντίκτυπο. Ο Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων θα θα, επίσης θα πρέπει να ε, συμμετέχει και να εξετάσει το πώς οι νέες προτάσεις θα συντεριαστούν επί τη βάση της δικής μου εμπειρίας θα έλεγα ότι όταν εγώ ήμουν Πρωθυπουργό. Δεν μου επαγόρευσε κανείς τι θα πρέπει να κάνω, αλλά αλλά υπήρχαν ε, φυσικά υποδείξεις για οικονομική σταθεροποίηση και, αλλά και οικονομικά κίνητρα δόθηκαν επί τη βάση ευρωπαϊκών κονδυλίων που υπήρχαν διαθέσιμα με τις συγκίσεις εξαγωγών καθώς και το τρίτο στοιχείο που μας επέτρεψε να μειωθεί η κοινωνική πίεση ήταν η επέκταση του δικτύου κοινωνικής πρόνοιας έτσι ώστε να ε, προστατευτούν οι ιδιαίτερα ευάλωτοι πληθυσμοί. Επόμενο ομιλητή, ο Στέβεν Βόλφ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης που ήρθατε σήμερα εδώ. Προτίμαζα διαφορετική ερώτηση και άκουσα την μία πρόταση που συνέδε ε, εσά, ε, την κυρία Βέστιγκερ, τον κύριο Χίλ και τον κύριο Μοσκοβισή. Και αυτό ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τεράστια επιτυχία. Είναι τεράστια επιτυχία, ότι έχει αντιμετωπίσει επιτυχώ την κρίση. Είμαι πραγματικά απογοητευμένο που υπάρχει κόσμο σε αυτή την αίθουσα που δεν αναγνωρίζει ότι η διάσωση του ευρώ στην ουσία σήμανε τη θυσία εκατομμυρίων ε, ζωών, ανθρώπων, αποταμιεύσεων αυτών για των ζωών του. Και έχω συναδέλφου εδώ δίπλα που συμφωνούν μαζί μου. Το θέμα δεν, το να σωθεί το ευρώ δεν σημαίνει να σωθεί η Ευρώπη. Η διάσωση του ευρώ σημαίνει κοινή τραπεζική πολιτική, κοινή δημοσιονομική πολιτική και συνεχής βούληση για να υπάρχουν τεράστιες οικονομικές μεταφορές, ε, βάσματα από τις πλούσιες χώρες στις στοχές χώρες. Δεν βλέπετε ότι όταν το κάνετε αυτό αυτός ο βασικός λόγος για να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η Ευρώπη και να εξοικονομεί, να εισαιωθεί μάλλον το ευρώ, θα πρέπει η εθνική ανεξαρτησία να χαθεί και να χαθούν οι δημοκρατικές αξίες με απαράδεκτο τρόπο. Well, uh, uh, uh, uh Mr. Wolf, first of all, uh, Κύριε Βόλφ, πρέπει να σημειώσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν συμφωνώ με την ανάλυση σας και τον ρόλο που θεωρείτε ότι έχει παίξει το ευρώ στην οικονομία της ε, Ένωσης. Βεβαίω, ξέρω πως διαφορετικές χώρες ακολούθησαν διαφορετικές προσεγγίσεις, κάποιες άλλες έμειναν εκτός της Ευρωζώνης, αλλά θα αναφερθώ και πάλι στην εμπειρία της δικής μου χώρας. Το 2008-2009 περνούσαμε πολύ σοβαρή οικονομική κρίση χωρίς το ευρώ και άλλες χώρες επίσης το ίδιο. Οπότε το ευρώ δεν είναι ε, το βασικό πρόβλημα εδώ πέρα. Εάν αντιμετωπίζουμε οικονομική και κοινωνική κρίση στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κρίσης και ε, νομίζω ότι τουλάχιστον την παγκόσμια κρίση δεν τη δημιούργησε το ευρώ, τότε οι χώρες εκείνες οι οποίες είχαν κάποιες αδυναμίες επηρεάστηκαν από αυτή την κρίση και πράγματι δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο για να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Όχι τέλειο, κανείς δεν λέει κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο να βοηθηθούν αυτές οι χώρες και πράγματι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο, να φροντίσουμε να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα δημοσιονομικά μεγέθη αλλά και την κοινωνική διάσταση και πολλές από τις ε, προκλήσεις που αναφέρατε εγώ θεωρώ ότι αντιμετωπίζονται μόνο αν συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ζαριανόπουλος κατόπιν. Κύριε Ντομπρόφσκι, σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσει σε όλους τους τόνους ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και τα Μνημόνια Διαρκείας ισχύουν απαρέγκλητα, ανεξάρτητα από το μείγμα διαχείρισης, περιοριστικό ή επεκτατικό. Η Ένωση γνωρίζοντας ότι τα αντιλαϊκά μέτρα αλλά και οι αγώνες εναντίον τους θα κλιμακωθούν, ήδη συζητά για τον περιορισμό, δηλαδή την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, όπως με την πρόταση Μόντι, ή όπως χαρακτηριστικά κάνει αυτό τον καιρό μέσω της Τρόικα στην Ελλάδα με απέτηση κατάργησης του δικαιώματος απεργίας από εργοδότες και με τη συμφωνία της κυβέρνησης. Τελικά, ο κοινωνικός διάλογος που πάντα καταλήγει σε συρρήκνωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, σε τι άλλο χρησιμεύει πέρα από την ομιμοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Μάλιστα, θα το πω αγγλικά. Όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, υπάρχει μια σαφής δέσμευση του Προεδρού Γιούνκερ και της νέας Επιτροπής για να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευελιξία στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου σταθερότητας, κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε. Και υπάρχει εδώ πέρα ε, η δυνατότητα για σταθερότητα και με μέτρα προληπτικά και ε, διορθωτικά και ε, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και τι χρειάζεται να κάνουμε, χρειάζεται να εφαρμόσουμε αυτή την ευελιξία. Όσον αφορά το δικαίωμα στην απεργία και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα. Είναι σαφές πως ε, είναι κομμάτι αναπόσπαστο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και έτσι πρέπει να παραμείνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κάρινς από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντομπρόφσκης, τον Ιανουάριο φέτος η Λετωνία μπήκε στην ε, Ευρωζώνη και σε λίγους μήνες θα μπει και η Λιθουανία. Ταυτόχρονα ακούσαμε να λέγεται πως ε, μαζί με την ένταξη στην Ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να μην γίνει άλλη διεύρυνση. Κάποιες ερωτήσεις λοιπόν. Πώς αξιολογείτε εσείς την ένταξη της Λετωνίας και την προσεχή ένταξη της Λιθουανίας. Και δεύτερον, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να σταματήσει η διεύρυνση της Ευρωζώνης και ανέγεται. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρινς για την ερώτηση. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ένταξη της Λιθουανίας, ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό η ίδια ανάλυση με την ε, Λετωνία. Εγώ θεωρώ πως τα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομίσματα που ήταν ούτως ή άλλως συνδεδεμένα με το ευρώ, όπως το ΛΑΤ και το ΛΙΤΑΣ των δύο αυτών χωρών, ε, καλά θα κάνουν να ενταχθούν γιατί βεβαίως ε, έχουν την ασφάλεια ενός μεγάλου νομίσματος και γνωρίζουμε πως ε, υπάρχουν υπάρχει το κόστος το συναλλαγματικό το οποίο αποτρέπει συχνά τους επενδυτές μειώνονται επίσης τα επιτόκια και ε, ήδη ε, η Λετωνία εκμεταλλεύεται αυτά τα πλέον και βέβαια υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα. Αν δούμε το τι γίνεται με τη Ρωσία και την Ουκρανία και τις υπόλοιπες γειτονικές μας χώρες. Νομίζω πως ε, σε αυτή την περίπτωση η στενότερη ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το συμφέρον των χωρών μας. Τώρα όσον αφορά την περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωζώνης, η Ευρωζώνη πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και νομίζω θα διευρυνθεί, αλλά πέρα από την ε, Λιθουανία και την ε, Δανία, ε, οφείλουμε να πούμε πως δεν υπάρχει άλλη χώρα με τους απαραίτητους δεσμούς. Και αυτή τη στιγμή κανένας άλλος δεν θέλει να ενταχθεί στο ευρώ, έτσι. Και Εντάξει, υπάρχουν άλλες χώρες ε, ε, οι οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Σας ευχαριστώ, Ρενάτο Σόρου, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, ναι. Άκουσα να λέτε κάποια σωστά πράγματα σε σχέση με το γεγονός ότι στην Ευρωζώνη θα πρέπει να δεσμευτούμε όχι μόνο στη σύγκληση των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών αλλά και στη σύγκληση των κοινωνικών πολιτικών. Δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την Ευρωζώνη αν δεν καταφέρουμε να φέρουμε κοντά και τις κοινωνικές ε, πολιτικές των διαφορών χωρών. Ταυτόχρονα όμως σας άκουσα να λέτε με περηφάνεια το πόσα έγιναν στη χώρα σας ε, και που τους επόμενους μήνες ε, θα μπει επιτέλους στην Ευρωζώνη. Δεν μας είπατε όμως τίποτα για το τι έγινε στα επίπεδα φτώχεια της χώρας σας, πόσα στερήθηκαν, πόσο σοβαρά στερήθηκαν ε, πάνω από 63% αυξήθηκε η ηλική στέρηση στη χώρα σας. Δεν μας είπατε τίποτα γι' αυτό, Τι για τα επίπεδα ανεργίας, τα οποία κάθετα ε, υψώθηκαν και μόνο πρόσφατα άρχισαν κάπως να κάμπτονται. Ο συνάδελφος Σάιμον πριν από λίγο είπε ότι όντως κάνατε λάθη. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα λάθη που πιστεύετε ότι κάνατε και ποια είναι τα λάθη που δεν θα επαναλάβετε πια στην ενδεχόμενη νέα θέση σας. Θα μπορούσατε επίσης να μου πείτε, συνάδελφε, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος και διακόπτη. Ο κύριος Δομπρόφσκης. Ε, Σε σχέση με την εμπειρία της ε, Λετωνίας και τα προβλήματά της, θα ήθελα να πω ε, Η χώρα μας πέρασε μια μεγάλη οικονομική και δημοσιονομική κρίση, η οποία ήταν ήδη ε, βαθύτατη και ήταν ε, ήδη σε ένα πρόγραμμα δανεισμού η λετονία Λετωνία όταν αναλάβαμε εμείς ε, την κυβέρνηση με αποστολή ακριβώς να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία βεβαίως ε, προέκυψαν ε, στη θητεία της ε, προηγούμενης κυβέρνησης. Και όπως είπατε πράγματι η δικιά μας δουλειά ήταν να δημιουργήσουμε οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας το συντομότερο δυνατόν. Κάτι το οποίο έγινε. Και βεβαίως όταν ε, το κράτος αντιμετωπίζει τέτοια κρίση, δηλαδή 14% μείωση του ΑΕΠ, ε, δεν είναι δυνατόν βεβαίως να την ξεπεράσει χωρίς ε, συνέπειες. Το θέμα είναι μετά πώς θα την ξεπεράσει και πόσο γρήγορα. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν και τονίσαμε τρεις πτυχές. Η κοινωνική πτυχή παρά τα μέτρα λιτότητας ε, υπήρχε ένα κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας, ένα επιπλέον μάλιστα ακριβώς για τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από την κρίση. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα ήταν ε, δημιουργία θέσεων εργασίας και υποστήριξη ατόμων που δούλευαν ε, part-time, πρόσβαση στα φάρμακα, και στήριξη διαφόρων ευπαθών ομάδων. Σας ευχαριστώ. Μπέντ Λούκε από το ECR. Κύριε Ντομπρόφσκης, είπατε πως το ευρώ είναι μια επιτυχία και δεν φταίει για την ανεργία στην Ευρωζώνη. Πριν από μερικές εβδομάδες ε, στο Λίνταου συναντήθηκαν κάποιοι ε, νομπελίστες οικονομικών. Κρίστοφερ Σίμς και ο Πίτερ Ντάιμοντ και άλλοι είπαν πως η Ευρωζώνη δεν θα μπορέσει να ανακάμψει αν συνεχίσει να υπάρχει το ευρώ. Εσείς θα πείτε πως ξέρετε καλύτερα και δεν πρέπει να υπερτιμούμε το τι σημαίνει βραβείο Νόμπελ. Τι θα γίνει όμως εάν έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή θα μπορούσε μια χώρα να ε, θέλει να βγει από το ευρώ εάν ζήσει μια παρατεταμένη φάση ανεργίας και ύφεσης. Θα ε, φροντίσετε να το καταστήσετε νομικά δυνατόν να μπορέσει να αποχωρήσει δηλαδή μια χώρα εάν το θέλει και αν η απάντησή σας είναι όχι θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο δικαίωμα θα ε, εμποδίσετε εσείς μια χώρα που θα θέλει να αποχωρήσει από το ευρώ. Μάλιστα. για το ευρώ. Και την τάση αυτή που υπάρχει ε, για να κατηγορούμε το ευρώ για πράγματα που ξεκίνησαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Την απάντησα ήδη αυτή την ερώτηση πολλές φορές. Ε, εντάξει, ωραία. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος για τη συνθήκη. Γνωρίζουμε πως όταν συζητήθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας υπήρχε μια παρόμοια συζήτηση για το δικαίωμα των κρατών μελών να φύγουν από την Ένωση, κάτι το οποίο επίσης δεν ήταν δυνατόν στο παρελθόν. Οπότε, τελικά υπάρχει αυτό το δικαίωμα στη συνθήκη και έχετε δίκιο, πράγματι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται η δυνατότητα ενός κράτους μέλους να φύγει από το ευρώ ε, αν δεν φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα. Οπότε, ε, οπωσδήποτε η πρόθεση της Κομισιόν δεν είναι να καταθέσει μια τέτοια πρόταση, αλλά εάν υπάρξει μια αλλαγή της συνθήκης και τα κράτη-μέλη ζητήσουν μια τέτοια διάταξη, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούν, μπορούν να συζητήσουν τα κράτη-μέλη. Εξάλλου τα κράτη-μέλη ε, κυρώνουν τη συνθήκη. Εάν το επιθυμούν, μπορούν να βάλουν μια τέτοια διάταξη και έτσι ε, οπωσδήποτε αν υπάρξει αίτημα από τα κράτη-μέλη η Κομισιόν θα δώσει την τεχνική στήριξη που απαιτείται. Αλλά δεν είναι αυτή η πολιτική της Κομισιόν. Εσείς προσωπικά είστε υπέρ. Όπως σας είπα, εάν ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, η Κομισιόν θα δώσει την τεχνική στήριξη. In ε, εν πάση περιπτώσει χρειάζεται ομοφωνία για να τροποποιηθεί η συνθήκη. Νίλ Τόρβαρτς, από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ και σας ε, καλωσορίζω κύριε Ντομπρόφσκι, μιλήσατε για τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως στην περίπτωση της Λετωνίας ε, μιλήσατε για το δημοσιονομικό ε, σύμφωνο, για το 2-pack, για το 6-pack, για το μέσο σταθερότητας και ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως ε, να θέσουμε στην ε, κύρια οδό ε, αυτά τα, τα σύμφωνα. Όμως αυτό μπορεί να είναι και αμφίδρομο. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα, θα θέσετε αυτά τα μέσα και θα τα τοποθετήσετε ως κυρίαρχο ρεύμα. Όπως ξέρετε, θα πρέπει η νομοθεσία η ίδια να προβλέψει την αναθεώρηση του Six pack και του ΤΟΥΠΑΚ pack μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Και αυτό που έχει σημασία είναι να προβούμε σε μία αναθεώρηση προς τα πίσω, δηλαδή να δούμε ε, πώς λειτουργήσαν αυτά τα νομοθετήματα εξ αρχής, τον πρώτο χρόνο και μετά να δούμε πώς διαμορφώνονται οι αλλαγές πολιτικής. Δηλαδή μετά την πρώτη αναθεώρηση θα πρέπει να αναλύσουμε περαιτέρω. Τώρα, ως προς το, το κυρίαρχο αυτό ρεύμα, όπως σας είπα, μέσα στα πλαίσια της μακροοικονομικής διακυβέρνησης η διαδικασία αυτή είναι πολύ δύσκολη και είναι δύσκολο να εξηγηθεί στους πολίτες. Υπάρχει το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας μέσα στα πλαίσια της πρόληψης ή της αντιμετώπισης. Έχουμε τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, έχουμε την ε, διαδικασία ε, μακροοικονομικών ανισοτήτων με το, το σκέλος της πρόληψης και το σκέλος της αντιμετώπισης. Επίσης προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όχι μόνο το υπερβολικό έλλειμμα, αλλά και το υπερβολικό ε, χρέος, διότι θα πρέπει να δούμε πώς ε, πληρούν τα κράτη-μέλη τις προϋποθέσεις αυτών των εποπτικών μηχανισμών. Γιατί ίσως ε, ορισμένα στοιχεία μπορούν να τεθούν υπόψη των κρατών μελών, δηλαδή εκεί που υπάρχουν διαφοροποιήσεις, γιατί πολλές φορές ε, υπάρχει και σύγχυση μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη. Γκουε. Ευχαριστώ. Όλοι αναγνώρισαν ότι η στρατηγική της Λισαμπόνας ήταν μια αποτυχία. Η Ευρώπη 2020 δεν επιτρέπει τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας. Δεν υπάρχει καμία καινοτομία. Επίσης, το πρόγραμμα ανάκαμψης του Ιουνίου 2012 δεν απέδωσε καθόλου. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε άρδιν τις πολιτικές μας βγαίνοντα από τη λιτότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια και ανθρωπιστικά καθώς και περιβαλλοντικά. Αντί να μιλάμε μόνο για νομισματικό ανταγωνισμό, το ευρώ δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα μέσο συνεργασίας έτσι ώστε να προωθήσουμε την, ε, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σε σχέση με το θέμα αυτό τη στρατηγική της Λισαβόνας και της Ευρώπης 2020 ξέρουμε ότι θα βασιστούμε στην αναθεώρηση της Ευρώπης 2020 γιατί όταν συντάχθηκε αυτό το πρόγραμμα ε, αυτό έγινε πριν ανακύψει η κρίση της Ευρωζώνης. Γι' αυτό στην αναθεώρηση θα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διδάγματα της κρίσης, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Αυτό είναι απόλυτα σαφές και θα πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης της Ευρώπης του 2020 αναφέρατε. Επίσης και τα περιβαλλοντικά ε, μέτρα. Εάν δείτε την, ε, το πρόγραμμα Ευρώπη 2020, έχουμε περιβαλλοντικούς στόχους και βρισκόμαστε πολύ κοντά στα τελικά αποτελέσματα. Όμως ε, θα πρέπει να οικοδομήσουμε αυτό το πλαίσιο πέρα από την Ευρώπη 2020 σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι άλλοι δείκτες είναι καθαρά ενδεικτικοί, ενώ οι ενεργειακοί δείκτες, μείωση των εκπομπών, οι λεγόμενοι στόχοι 20-20-20 είναι δεσμευτικοί προς τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη πρέπει να τους εφαρμόσουν. Ως προς την Ευρωζώνη ως μέσο για επενδύσεις αναφέρομαι σε αυτή την πρόταση των 30 δις αυτού του πακέτου το οποίο θα πρέπει να ισχύσει τα επόμενα τρία χρόνια. Σας ευχαριστώ. Είμαστε στο ίμιση τώρα της ακροασής μας και θα δώσω την προεδρία στη συνάδελφο Μαρίτα Ούλσκβοκ εξ ονόματος της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην Μόνικα Βαβάνερ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε Επίτροπε. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο θέμα της δημοκρατικής νομοποίησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το θέμα της διοργανικής συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο δεν έχει κάποιο ρόλο στην εποπτεία αυτού του ζητήματος και ακόμα και οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου αγνοούνται από το Συμβούλιο. Θα φροντίσετε να προταθεί μια διοργανική συμφωνία για να εκπληρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ρόλο του στην έγκριση ετήσιας έκθεσης και κατευθυντηρίων γραμμών και δεύτερον η κοινωνία των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Μας είχε υποσχεθεί κατευθυντήριες γραμμές ήδη η προηγούμενη Κομισιόν για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Γιούνκερ, πρότεινε να το κάνει αυτό. Πότε ακριβώς λοιπόν θα δούμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προτείνετε εσείς γι' αυτό, ειδικά δεδομένων των ε, προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, ε, για την διοργανική συμφωνία. Νομίζω πρώτα απ' όλα πως πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία. Να δούμε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά για να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και με τα άλλα θεσμικά όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις και πραγματικά να ε, επικεντρωθούμε στην ουσία στο τι είμαστε διατεθειμένοι να επιτύχουμε και ως ε, Ευρωβουλευτής και εγώ είμαι διατεθειμένος να εργαστώ προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε ε, ουσιαστικά αποτελέσματα. Για την συμφωνία πλαίσιο. Θα πρέπει, αν θα πρέπει να γίνει στο υφιστάμενο πλαίσιο που υπάρχει ή αν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε όταν συμφωνήσουμε επί της ουσίας, δηλαδή το πώς και το που ακριβώς θα διασφαλίσουμε αυτή τη συνεισφορά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τώρα για τους κοινωνικούς εταίρους. Ήδη ανέφερα κάποιες ιδέες και Νομίζω αυτές θα τις αναπτύξουμε περαιτέρω με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά περιθώριο για περαιτέρω εμπλοκή τους στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη και στο εθνικό επίπεδο, στην εις εξέταση, νομίζω μπορεί να γίνει, όπως και στην προετοιμασία των χωρών, των συστάσεων αναχώρα. Ο κύριος Τσάνη. Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Λούκ πριν από λίγο για την έλλειψη της νομοθετικής ψήφου που υπάρχει για να πετρέψει σε κάποια από το ευρώ. Θα ήθελα να σταθώ στα εξή. Πρώτον, όσον αφορά την είσοδο στο ευρώ, οι αποκλήσει ε, νομοθεσίας που υπάρχουν στις διάφορες χώρες είναι σημαντικές. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία έχουν συμφωνίες που τους επιτρέπουν να μην εισέλθουν στο ενιαίο νόμισμα, ενώ όλες τις άλλε χώρε που δεν είναι στο ευρώ πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια σύγκλησης για να μπουν. Αυτό την πρώτη γνώμη που σας ζητώ είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι στο εξή που είπατε ότι όσον αφορά μια νομοθεσία για την έξοδο από το ευρώ, αυτό θα πρέπει να απασχολήσει το Συμβουλίο, όμως στις 25 Μαΐου οι Ευρωπαίοι πολίτες έδωσαν σαφή εντολή. Δεκάδες εκατομμύρια ψήφισαν κόμματα που ζητούσαν την έξοδο από το ευρώ στο δημοψήφισμα για το ευρώ. Εσείς θα αποφασίσετε να αγνοήσετε αυτή τη φωνή και να περάσετε τον μπαλάκι στο Συμβούλιο ή θα κάνετε κάτι ώστε να πιέσετε το Συμβούλιο για να φτάσει να ασχοληθεί με τέτοιου είδους νομοθεσία. Να θυμίσω ότι η μεταρρύθμιση της ΟΝΕ είναι ανάμεσα στις 10 προτεραιότητες που ενέφερε ο Πρόεδρος Γιούγκερ. Άρα είναι προτεραιότητα για όλους. Θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας. Κύριε Ντομπρόφσκη, έχετε το λόγο. Όσον αφορά τα διάφορα σενάρια για τα διά, και διαφορετικές ε, ρυθμίσεις για τα διάφορα κατεμέλη. Ξέρουμε ότι η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιλέξει να μείνουν εκτός. Είναι κάτι το οποίο επέλεξαν ε, κατά τη δημιουργία της Ευρωζώνης. Αλλά για τα μη κρατημέλη που μπαίνουν το 2004 και μετά δεν έχει προβλεφθεί ε, το opt-out. Δεν Δεν είναι μόνο μια επιλογή, αλλά είναι υποχρέωση των νέων κρατών μελών να μπουν στο ευρώ στην Ευρωζώνη από τη στιγμή που θα πληρούν τα κριτήρια του Μάστριχτ. Αλλά γνωρίζουμε ότι διάφορα νέα κρατημέλη έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε όλα αυτά. Τα περισσότερα έχουν ήδη μπει στην Ευρωζώνη. Ορισμένες χώρες ιδιαίτερα με κειμενόμενα συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν είναι μέσα στον ε, μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμίων γιατί σημαίνει μεγάλες αλλαγές νομισματικής πολιτικής πρέπει να οριστούν για να σταθεροποιηθούν τα οι συναλλαγματικές τους ισοτιμίες και πρέπει να σκεφτούμε ένα μέσο για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε αυτές τις οικονομίες. Αν κάποιες χώρες βασίζονταν σε αυτό το μέσο, πρόκειται για μεγάλη και σοβαρή πολιτική αλλαγή. Όσον αφορά την αλλαγή συνθήκης και τις δυνατότητες για τις χώρες της Ευρωζώνης να φεύγουν από την Ευρωζώνη, όπως ήδη ανέφερα, αυτό είναι κάτι που καταρχήν πρέπει να απασχολήσει και τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ένωσης και να ζητήσουν μέσα στο πλαίσιο των λαγών των συνθήκων, όπως είναι και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και όπως είναι και με τη δυνατότητα να εγκαταλείψει κανείς την Ένωση. Αλλά βέβαια όχι. Δεν είναι μια κατεύθυνση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, την υποστήριξει δραστήρια ή θα την ενθαρρύνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μάρκος Φέρμπερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Στον τομέα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ποιες είναι οι προτάσεις σας για το πόσο μπορεί να δοθεί περισσότερο βάρο στις συστάσεις αναχώρα και το τι μπορεί να γίνει επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ειδικά όσον αφορά τον λεγόμενο νόμο περί μικρών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Okay. Ε, ε, thank you, ε, Mr. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Φέρμπερ. Καταρχήν όλες οι ειδικέ συστάσεις για την αναχώρα Όντως πρέπει να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή αυτών των συστάσεων δεν ε, είναι τόσο στενάριο όσο θέλαμε. Διάφορες εκτιμήσεις ε, τοποθετούν στο 10 με 40%. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αποτιμά στο 18%. Πάντως είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν ε, κυρώσεις ε, οι οποίες να συνοδεύουν αυτές τις συστάσεις αναχώρα. χώρα. Ούτε αυτή είναι η πρόθεσή μας. Η ιδέα εδώ είναι στην ουσία να ενισχύσουμε την ιδιοποίηση των συστάσεων αυτών αναχώρα. Δηλαδή πραγματικά να συζητήσουμε πιο εις βάθος με κάθε κράτος μέλος και τους κοινωνικούς εταίρους της χώρας για αυτές τις συστάσεις. Επίσης, ε, να συζητήσουμε τη χρηματοδότηση από την Ένωση, λειτουργικά προγράμματα, ώστε να εξασφαλίσουμε πράγματι ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα γίνεται ε, σε συμφωνία με τις ε, αναχώρας συστάσεις, έτσι ώστε να ισχύσουν και οι όροι, η αιρεσιμότητα για τις συστάσεις αυτές και τη χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα δεύτερο γύρο θα μπορέσει να είναι πιο συγκεκριμένη όσον αφορά τις τη θέσεις και να δώσει και στόχους. Τώρα, εάν δεν συμμορφωθούν αυτές οι χώρες και έτσι οδηγηθούν σε εξαιρετικές ανισορροπίες, όπως ε, με την ε, διαδικασία υπερβολικού χρέους, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχες διαδικασίες. Α, με συγχωρείτε, ναι. Νομίζω πως τη δεύτερη πρέπει να την απαντήσω διμερώς ή αν υπάρξει κάποια επερώτηση, γιατί δεν έχω χρόνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερνάντες του, των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Ντομπρόφσκης. Όλοι συμμεριζόμαστε την έννοια ενός κοινού νομίσματος ε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χώρες που έχουν μεγάλο χρέος μπορούν να ακολουθήσουν πορεία free rider. Γι' αυτό υπάρχει και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Επίσης υπάρχει και η στάση free rider εκείνων οι οποίοι έχουν, πολύ, ε, έχουν υπερβολικό χρέος και δεν μπορούν να υποτιμήσουν ε, το νόμισμά τους κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ε, μέτρα τα οποία προέρχονται από το, το πλεόνασμα αλλά και από τα ελλείμματα. Αυτό που πρέπει λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε είναι και το έλλειμμα αλλά και το πλεόνασμα του τρεχούμενου, των τρεχούμενων λογαριασμών. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν ειδικέ συστάσεις ανακράτος και θεωρείτε ότι οι, οι, οι χώρες οι οποίες έχουν ε, πολύ υψηλό πλεόνασμα θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή αντιμετώπιση μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Απάντηση. Άρα το βασικό ερώτημα αφορά ε, το ισοζύγιο τρέχουσων ε, λογαριασμών, τα ελλείμματα και το πλεόνασμα. Και φυσικά τα μεγάλα ελλείμματα δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα ανταγωνισμού εξαγωγών, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και είναι ένας δείκτης ο οποίος θα δημιουργήσει ανησυχίες για την εν λόγω χώρα. Βέβαια το έλλειμμα σε μία χώρα σημαίνει πλεόνασμα σε μία άλλη. Γιατί ο, θα πρέπει να υπάρξει εξισορροπημένος ισολογισμός. Γι' αυτό καθίσταται σαφές ότι το ζήτημα αυτό το οποίο συζητούν οι ΕΚΤ και οι οικονομολόγοι θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ε, ζήτηση στις πλεονασματικές χώρες. Αυτό είναι το ένα σκέλος της, εξίσωσης και θα πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές, δηλαδή τις ελληματικές χώρες αλλά και τις ε, πλεονασματικές, για να δούμε τι μπορεί να γίνει για να δώσουμε ειδική όθηση στη ζήτηση, ιδιαίτερα στις ε, πλεονασματικές ε, χώρες, διότι αυτές οι δύο έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. ολουρίκε Τρεμπέσιους από το ECR. Εδώ είμαι, κύριε Ντομπρόφσκης. Θεωρείστε ως πρώην Πρωθυπουργός της Λετωνίας ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος επέβαλε σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην χώρα του. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω στο πλαίσιο αυτό εάν είστε υπέρ μιας ευρωπαϊκής ε, πολιτικής για την ανεργία. Μήπως με αυτόν τον τρόπο απλά μεταθέτουμε στο πρόβλημα τα ουσιαστικά και διαρθρωτικά προβλήματα και εδρεώνουμε την ανεργία και μήπως έτσι τιμωρούνται χώρες όπως η Γερμανία η οποία έχει ευέλικτη ε, αγορά εργασίας ή χώρες όπως η Λετωνία που έκανε τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις τι σκοπεύετε να κάνετε για να προωθήσετε και να επιτηρήσετε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο μέλλον και τέλος ποιους άλλους μηχανισμούς μεταφοράς χρημάτων σκοπεύετε να εισαγάγετε ή να ενισχύσετε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή που αφορά μια κοινή πολιτική και πιθανώς ε, ασφάλιση ή επίδομα για τους ανέργους. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία βεβαίως σχετίζεται και με την φοροδοτική ικανότητα της Ευρωζώνης, αλλά επίσης πρέπει να πούμε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνένεση για κάτι τέτοιο στο Συμβούλιο και οπωσδήποτε αν θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε αλλαγή της συνθήκης. Χωρίς αλλαγή της συνθήκης δεν γίνεται. Και επίσης ε, είναι σαφές πως ε, περισσότερη αλληλεγγύη σημαίνει και περισσότερος έλεγχος και περισσότερη ευθύνη. Αυτά πάνε μαζί. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν τίθεται το ζήτημα τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον. Ίσως με κάποια αλλαγή της συνθήκης ε, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αλλά αυτό το οποίο θα κάνει και θέλει να κάνει η νέα Επιτροπή είναι να διασφαλίσει πως τα επιδόματα της ανεργίας στα διάφορα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούνται στόχευμένα και να αφορούν ακριβώς τους νέους που είναι και τις διάφορες ομάδες που είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Ειδικά για τους νέους έχουμε την ε, πρωτοβουλία την σχετική και βεβαίως και παραδείγματο χάρη τους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν φτάσει ακόμα στην ηλικία συνταξιοδότησης. Οπότε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εργαστούν τα κράτη-μέλη πιο στοχευμένα. Για να του από τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, η Μαριάν Τάισεν σε πέντε φορές αναφέρθηκε σε κοινωνικούς δείκτες στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και είπε πως είναι η φτωχή συγγενής και πρέπει να ενισχυθούν. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επίσης μίλησε για ενίσχυση της οικονομικής πτυχής στη χάραξη της ε, οικονομικής ε, πολιτικής. Δεδομένης της σχέσης σας και με τους δύο αυτούς, ε, ποια είναι η άποψή σας για την ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών δικτών και δεδομένων των προσφάτων σχολείων από κάποια κράτη-μέλη πως ε, μάλλον δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στο προτινόμενο χρονοδιάγραμμα. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει. Σε σχέση με τους κοινωνικούς ε, δείκτες, ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και με την ε, υποψήφια επίτροπο Τάισεν ότι οι δείκτες αυτοί πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχα επαναλάβει αρκετές φορές εδώ και θα ήθελα να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Γιούνκερ και την Επίτροπο Τάισεν έτσι ώστε να ενισχύσουμε την κοινωνική αυτή διάσταση και τους εν λόγω έτσι ώστε οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές να συμβαδίζουν με την κοινωνική πολιτική καθώς και την πολιτική απασχόλησης σε σχέση με την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Η ιδέα που πρέπει να μας διέπει είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών χρησιμοποιώντας την σχετική ευελιξία μέσα στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά ομοιογενή τρόπο, έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να την χάνουν ίσης μεταχείρισης. Αυτή είναι η γενική ιδέα και πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, να συνειδητοποιούν την συλλογιστική γιατί δηλαδή η πολιτική ευελιξία επιβάλλεται. Η Κωνσταντίνκα Κούνεβα, Κούνεβα, από την ε, ΓΟΕ. Είσαι σημασία στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Ωστόσο, στις χώρες που εφαρμόζονται προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής καταργούνται πολλά δικαιώματα, ακόμα και αυτό της απεργίας. Θα ήθελα να μου απαντήσετε με ένα ναι ή όχι, αν συμφωνείτε με την πίεση που ασκεί σήμερα η Τρόικα στην Ελλάδα να επιβληθεί ξανά το δικαιώμα της ανταπεργίας των εργοδοτών, το γνωστό lockout. Και αν δεν συμφωνείτε, πώς θα το αντιμετωπίσετε ως αρμόδιος για θέματα κοινωνικού διαλόγου. Μη μου μιλήσετε για τις εθνικές ε, ευθύνε των κρατών μελών. Θα ήθελα να ακούσω εσείς τι θα, τελέσετε, τι θα τελέσετε, να κάνετε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως μια πολύ σημαντική προτεραιότητα τη μείωση της στόχιας ως το 2020. Ως επίτροπος με κοινωνικές αρμοδιότητες που συνδέονται με το ευρώ, είστε έτοιμος να στηρίξετε ένα μεγάλο ρεύμα ευρωβουλευτών και ευρωπαίων πολιτών, ένα ρεύμα που ζητά από τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια με την ίδια αυστηρότητα όπως το έλλειμμα και το κρέος. Είστε έτοιμοι. Η πρόεδρος διεκόπτη την ε, κυρία Κούνεβα. Ο υποψήφιος επίτροπος, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καταρχήν, να πω και πάλι ότι όσον αφορά τις χώρες που είναι σε πρόγραμμα, το πρώτο βήμα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις της Τρόικα όχι μόνο εξετάζονται όσον αφορά τον οικονομική και δημοσιονομική τους ε, επιρροή, αλλά και όσον αφορά ε, την κοινωνική τους, ε, το κοινωνικό τους αντίκτυπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο βεβαίως είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε και να προβλέψουμε συγκεκριμένους μηχανισμούς για το πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό. Αναφέρατε δε κάποια συγκεκριμένα αιτήματα της ε, Τρόικα προς την Ελλάδα για τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω αλλά ε, σαφώς Είμαι πρόθυμος να το συζητήσουμε διμερώς από τη στιγμή που θα έχω εξοικειωθεί με περισσότερες λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις της Τρόικα στα διάφορα κράτη-μέλη. Και βεβαίως ως Αντιπρόεδρος για το Ευρώ και το Κοινωνικό Διάλογο σκοπεύω να συνεργαστώ πολύ στενά με τα κράτη-μέλη, με την Τρόικα αλλά και να προωθήσω την προτεραιότητα αυτή της Κομισιόν ώστε να είναι πολύ πιο σαφής η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου στην λήψη αποφάσεων. Σας ευχαριστώ. από τους Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις απαντήσεις σας μέχρι τώρα κύριε Ντομπρόφσκης βεβαίως. Καμιά φορά λέτε πως είναι δύσκολο να περάσει μια θέση από το σώμα των επιτρόπων. Θέλουμε όμως να ακούσουμε τη δικιά σας θέση τώρα. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις και θέλω να ακούσω την δικιά σας την άποψη. Πρώτα απ' όλα η σημασία των κοινωνικών δικτών. Τους αναφέρατε και σας ευχαριστώ. Αλλά το σημαντικό είναι εάν είστε διατεθειμένος να προχωρήσετε σε διορθωτικές με συγχωρείτε, κινήσεις όταν δεν κάνουν κάτι τα κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη όταν υπάρχει υπερβολική ανισότητα σε ένα κράτος Θα έχουμε διορθωτική δράση. Δεύτερον, για το ευρώ. Ήσασταν κάπως ασαφείς. Αφήσατε ανοιχτή την δυνατότητα αποχώρησης από το ευρώ, κάτι το οποίο δημιουργεί ασάφεια. Θέλουμε να ακούσουμε από εσάς προσωπικά θα στηρίξετε το ευρώ και θα φροντίσετε όλες οι χώρες του ευρώ να παραμείνουν σε αυτό. Uh, Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας ε, για την σημασία των κοινωνικών δικτών, συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο είπε και η Μαριάν Τάισεν εδώ στην δική της ακρόαση ότι δηλαδή πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στους κοινωνικούς δείκτες όταν μιλάμε για τις συστάσεις αναχώρα. Και εδώ πέρα συμφωνώ πλήρως με τη Μαρία Τάισεν και θα στηρίξω τις πρωτοβουλίες της ε, ως προς αυτό. Μετά, για πιθανές κυρώσεις. Γνωρίζουμε πως οι συστάσεις χώρα δεν επιφέρουν κυρώσεις, δεν επισύρουν κυρώσεις. Το έχω ήδη απαντήσει αυτό. Οπότε, εάν υπάρχουν υπερβολικές ανισορροπίες, ε, υπάρχει η σχετική διαδικασία και πράγματι σε αυτήν πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην κοινωνική πτυχή. Τώρα για το ευρώ. Νομίζω ε, πως είπα σαφώς πως ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα ενθαρρύνει η Κομισιόν. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ε, οπωσδήποτε είμαι υπέρ του ευρώ, εγώ έκανα εκστρατεία στη Λετωνία κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης για να μπει η Λετωνία και εξήγησα ακριβώς σε δύσκολες συνθήκες γιατί πρέπει να μπει η χώρα μου στην Ευρωζώνη, γιατί το ευρώ είναι σταθερό νόμισμα, γιατί έχει ε, ένα μέλλον ε, θετικό η Ευρωζώνη και γιατί ε, ακριβώς είναι καλή ιδέα για τα κράτη-μέλη να μπουν στην Ευρωζώνη. Πάντα ήμουν σαφής ως προς αυτό και πίεζα προς αυτή κατεύθυνση. Λάουρα Άγκια από την e Ιευτή. Ευχαριστώ. Κύριε Ντομπρόφσκης, ας μιλήσουμε για τον κοινωνικό διάλογο, γιατί η θέση σας για το ευρώ είναι απόλυτα σαφής Ξέρετε ότι ο κοινωνικός ε, διάλογος ε, αφορά τους κοινωνικούς εταίρους που οφείλουν να συμμετάσχουν. Εγώ είμαι Ιταλίδα και προέρχομαι από την Ουμβρία. Στην Ουμβρία υπάρχει μία βιομηχανική μονάδα πάνω από 130 χρόνια που ανήκει στην κοινοπραξία Tyson που προέβη σε μεγάλες ε, περικοπές. Ε, αυτό σημαίνει ότι χίλια, χίλια άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα στους επόμενους μήνες. Επειδή μιλάμε για πολυνικό, ε, κοινωνικό, με διάλογο, πιστεύετε ότι θα, είσαστε, θα είμαστε ένας πραγματικός συνομιλητής ή θα εκπροσωπούμε δύο διαφορετικές πραγματικότητες ή θέλετε πραγματικά κάτι να κάνετε στον τομέα του κοινωνικού διαλόγου. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Ως προς τον κοινωνικό διάλογο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κοινωνικός διάλογος ε, γίνεται σε πολλά επίπεδα, σε εθνικό και κοινοτικό. Όσον αφορά το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινωνικών εταίρων και μεταξύ κοινωνικών εταίρων αφεαυτών. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι κοινωνικοί εταίροι δεν είχαν προβάλει κάποια μεμονωμένη πρόταση, ολιστική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή όχι τομεακή. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Και πολλοί κοινωνικοί εταίροι θέλουν να προωθήσουν αυτό το διάλογο σε εθνικό επίπεδο τώρα. Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό μπορεί να κάνει είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή των ε, εθνικών κοινωνικών εταίρων σε θέματα συγκεκριμένης αρμοδιότητας. Βεβαίως, όταν μιλάμε για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χώρες, η εθνική κοινωνική εταίρη και η κυβέρνηση θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ορίσει καλύτερα το πλαίσιο δημιουργίας θέσεων εργασίας έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προβληματικοί τομείς που, στους οποίους αναφερθήκατε, Γέρομ Λένερς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόσκηση, Είναι πολύ ενδιαφέρον να σας βλέπουμε εδώ γιατί είσαστε επιτυχής επιτυχημένος πρωθυπουργός της Λετωνίας και στα πλαίσια της ε, Ευρωζώνης. Πολλοί βέβαια λένε ότι το έργο σας δεν είναι και τόσο καλό. Εγώ θα ήθελα οι περισσότεροι να μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Μία από τις βασικές προκλήσεις για την ΟΝΕ είναι να βρει ένα τρόπο για να ανταποκριθεί στα ασυμμετρικά σοκ χωρίς ε, να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και θα ήθελα να μου πείτε τι σκέφτεστε η τρέχουσα επιτροπή σκέφτηκε να συμπεριλάβει τα ε, διάφορα ευεργετήματα, ιδιαίτερα το επίδομα ανεργίας, κάτι το οποίο δεν, θεωρείς, θεωρώ σωστό. Εσείς τι γνώμη έχετε. Απάντηση. Αυτό το θέμα των ε, ασύμε, ασύμετρων ε, κλειδονισμών είναι ένα θέμα που έχει οδηγήσει σε διχογνωμίες και οι θέσεις διαφέρουν. Όμως έχουν ή μπορούν να αναλυφθούν ορισμένες πρωτοβουλίες που μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα εκείνες τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Και ε, αυτό αφορά την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων, την εγγύηση για τους νέους, τα δύο αυτά μέσα, δηλαδή έτσι ώστε να διευρυνθούν αυτά τα προγράμματα και να παραταθούν είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία. Τώρα, ως προς τη διευκόλυνση των επενδύσεων, μιλήσαμε για το πακέτο των 300 δις, όμως θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πακέτο υποβοηθά την οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, ιδιαίτερα σε χώρες υποπρόγραμμα. Επίσης υπάρχουν τα ευρωπαϊκά ταμεία μέσα στα πλαίσια του μόνιμου μηχανισμού μεταφορών και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους ε, πόρους πιο στοχοθετημένα και να προβούμε και προσυστάσεις στα κράτη-μέλη. Επίσης να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Περβάνς Περές, συγγνώμη, σοσιαλιστές, είπατε ότι θα θέλατε το ευρώ να στεφθεί από επιτυχία. Εσείς θα μπορούσατε να δεχτείτε μία χώρα να βγει από το ευρώ. Θεωρείτε ότι τα μακροοικονομικά μέτρα θα οδηγούσαν, ε, οδήγησαν μάλλον σε 250.000 εξόδους από τη χώρα σας. Μιλώ για τους νέους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να απασχοληθούν στη χώρα σας. Μιλήσατε για την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας. Πέρα από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα ευελιξίας που δεν χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα από τους προκατόχους σας μέσα στα πλαίσια των ευθυνών σας. Μιλήσατε και για πολιτικά σφάλματα στη χώρα σας, υπό τη δική σας ευθύνη. Θα ήθελα να μας δώσετε ένα τέτοιο σφάλμα, ένα παράδειγμα τέτοιου πολιτικού σφάλματος υπό την Πρωθυπουργία σας. Απάντηση. Ευχαριστώ. Πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, τρεις ήταν οι ερωτήσεις. Ουσιαστικά μιλήσαμε για την... Ε, μιλήσατε για τη Λετωνία, γι' αυτό θα απαντήσω στη γλώσσα μου. Όσον αφορά λοιπόν την κρίση στη χώρα μου, εγώ ανέλαβα την ε, κυβέρνηση σε μια στιγμή στην οποία ήμασταν πραγματικά στη χειρότερη στιγμή της ε, κρίσης. Είχαμε μείον 14% ε, ύφεση και αναλάβαμε την κυβέρνηση με έναν απλό στόχο, να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη το συντομότερο δυνατόν. Μέσα σε ένα χρόνο καταλήξαμε σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Προωθήσαμε τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και με τα μέτρα αυτά καταφέραμε να ε, πάμε σε μια κατάσταση στην οποία η κατάσταση, η οικονομία με της Λετωνίας είναι μια από τις οικονομίες που αναπτύσσονται ταχύτερα στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να ε, λύνουμε τα προβλήματα, αλλά με τρόπο ενεργητικό. Τώρα, για το σύμφωνο σταθερότητας, πράγματι δεν φτάνει ο χρόνος, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μία κάποια ευελιξία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Βεβαίως, ε, μπορείτε να θέσετε, άμα θέλετε, άλλη μία ερώτηση, ερώτηση να απαντήσω ή να το δούμε διμερώς. κυρία Μάκιντάιρ από το ECR έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε, εδώ είμαι, εδώ. Κύριε Ντομπρόφσκης, όπως είπατε, γνωρίζετε πως ε, οι μηχανισμοί κοινωνικού διαλόγου στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους σε εθνικό επίπεδο. Οι κοινωνικοί εταίροι ε, θα έχουν ίσως το δικαίωμα να διαπραγματευτούν συλλογικές συμβάσεις ε, με πανευρωπαϊκή ισχύ. Και εάν γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί το Συμβούλιο να δεχτεί ή να απορρίψει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί να τις τροποποιήσει. Στη δε προηγούμενη ολομέλεια ε, περάσαμε μια έκθεση με τίτλο «Πώς θα δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις νέες επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας». Μεταξύ άλλων λοιπόν η έκθεση αυτή ζητούσε από τους κοινωνικούς εταίρους να χρησιμοποιήσουν έξυπνα εργαλεία για να μειωθεί ακριβώς ο αντίκτυπος τυχών αποτυχημένων συνομιλιών και να στέλνουν ε, τις λεπτομέρειες στο Συμβούλιο αξιολόγηση Κοινωνικού Αντικτύπου της Κομισιόν. Θα μπορούσατε λοιπόν να μου πείτε πώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα έξυπνα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Well, uh, thank you for this, uh, question. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όσον αφορά τους, uh, τις αυτόνομες συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, οπωσδήποτε είναι δικαίωμά τους να συνάψουν τέτοιες. Και οριζόντιες ε, και στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή κλαδικές συμφωνίες. Και οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή ε, υπάρξει μια τέτοια συμφωνία και ζητηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους να μεταφραστεί σε νομοθεσία, οπωσδήποτε η Κομισιόν θα ξεκινήσει τη σχετική εργασία. Αλλά οπωσδήποτε η αξιολόγηση αντικτύπου ε, των αυτόνομων αυτών συμφωνιών όπως και άλλων νομοθετικών προτάσεων πρέπει να γίνει και να καλύψει τις διαφορετικές ε, πτυχές ε, οικονομικές, κοινωνικές έτσι ώστε τελικά να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη πρόταση και ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα και οπωσδήποτε Είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ με την ε, κυρία Μαριάν Τάισεν, υποψήφια επίτροπο, για να δούμε την σχετική έκθεσή σας ε, και να δούμε πώς το σύστημα αυτό των αυτόνομων ε, συμφωνιών θα προχωρήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. τώρα από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση για τον κοινωνικό διάλογο. Μέχρι στιγμή είμαι πολύ ικανοποιημένη από τις απαντήσεις σας για τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα έγιναν στην ε, συζήτηση της Ολομέλης όταν ο υποψήφιος ε, τότε πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ελάχιστοι μισθοί σε όλα τα κράτη-μέλη και ότι θα προβεί σε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, σύμφωνα με τις συνθήκες και όπως ήδη είπατε κι εσείς, η μισθή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κύριε Ντομπρόφσκη, σε ποια μέτρα θα λάβετε εσείς ώστε να εξασφαλίσετε το κοινωνικό διάλογο και τι αρμοδιότητες των κοινωνικότερων αν η Κομισιόν αναλάβει πρωτοβουλίες σε σχέση με τα, τους ελάχιστους μισθούς. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά ελάχιστος μισθούς στα κράτη-μέλη. Είναι βέβαια η πρόταση του Προέδρου Γιούγκερ, με την οποία συμφωνώ. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλα τα κρατημέλη να θεσπίσουν μήνυμο μισθούς, ελάχιστος μισθούς. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε μέσω των συστάσεων αναχώρα και επίσης ε, σε διάλογο με τα, κράτη. Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, διαφορετικά μοντέλα κοινωνικού διαλόγου και ότι σε ορισμένε χώρες, ιδιαίτερα ας πούμε στις βαλτικές χώρες όπου υπάρχει πολύ ισχυρός ε, κοινωνικός διαλόγος, υπάρχει αυτή η τάση οι ελάχιστη μισθοί να ορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους. Βεβαίω δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι κατά των κοινωνικών εταίρων εφόσον υπάρχει συνένεση ανάμεσα σε αυτούς. Εν γέννη όμως η Ευρωπαϊκή Κομισιόν θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ελάχιστους μισθούς. Το λόγο έχει ο Έντουαρτ Κούκαν από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θυμάμαι μία από τις γραπτές σας απαντήσεις ε, στην οποία γράψατε ότι θα εθαρρύνετε τα κρατημέλη για να έχουν ε, πιο ανοιχτέ ε, αγορές εργασία που θα ανταποκρίνονται και θα, ε, στη ζήτηση και θα ε, περιλαμβάνουν όλους. Θέλω όμως να σα θυμίσω πως ο ευρωπαϊκός Πληθυσμό γυράσκει και πρέπει να εγγυηθούμε εκείνου που έχουν περάσει τα 50 και που είναι κοινωνικά και οικονομικά δραστηριοί ότι δεν θα υποστούν διακρίσεις στην αγορά εργασία. Πώ θα εξασφαλίσετε λοιπόν ότι αυτή η δράση σα θα λαμβάνει υπόψη τη γύρανση του πληθυσμού και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε την ε, πραγματική συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην μελλοντική σας ε, εργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Κούκαν για τις αγορές εργασίας και τη γύραση του πληθυσμού. Είναι ένα, μία από τις βασικές προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο, διότι είναι σαφές ότι είναι πιο εύκολο να στηριχθεί ένα κοινωνικό πρότυπο όταν αυξάνεται ο πληθυσμός ή όταν είναι σταθεροποιημένες οι ηλικιακέ δομές, παρότι με έναν γυράσκοντα πληθυσμό. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς θα προσαρμόσουμε τα κοινωνικά μας συστήματα και τα συστήματα απασχόλησης ώστε να ε, συμβαδίσουν με την γυράσκουσα πραγματικότητα της Ευρώπης. Είναι πραγματικά σημαντικό να προωθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μείνουν στην αγορά εργασία, αν μπορούν, και επίσης να παρέχουμε στοχοθετημένη βοήθεια σε εκείνους οι οποίοι έχουν φτάσει στην ηλικία ταξιδότησης και που συχνά έχουν δυσκολία να βρουν ε, κάποια... είναι κοντά στις ηλικία μάλλον και δεν μπορούν να βρουν εύκολα δουλειά. Θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν μια νέα κατάρτιση επί τη βάση των... της ζήτησης της αγοράς εργασίας ώστε να μπορέσουν πραγματικά να μείνουν δραστήριοι ενεργοί όσο γίνεται περισσότερο. Ε, όμως είναι σοβαρή αυτή η πρόκληση και μας απασχολεί εδώ και χρόνια και πρέπει όλοι μαζί να αναζητήσουμε μια κατάλληλη απάντηση. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο, στην κυρία, με συγχωρείτε, Στάινρακ. Κύριε Ντομπρόφσκης, μία ερώτηση πρώτα απ' όλα για αυτά τα οποία είπατε για την οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων. Δεν ξέρω τι εννοούσατε εκεί πέρα ακριβώς ε, ίσως να έφταγε η διερμηνία μετά η κυρία Τάισον μας υποσχέθηκε πως θα έχουν ίσο ρόλο οι κοινωνικοί δείκτη, δείκτες στο ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο εσείς μιλήσατε για μια κάποια ενίσχυσή τους ε, ποιος έχει δίκιο τελικά μετά η Κομισιόν κατέληξε σε μια οδηγία για τον κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο των κομωτών, των οποίων όμως μετά δεν προωθήσατε στο Συμβούλιο. Πότε θα προωθήσετε αυτή την οδηγία πλαίσιο στο Συμβούλιο. Okay, uh, Ευχαριστούμε κυρία Στάινμπρουκ. Τρεις ερωτήσεις έχετε υποβάλει σε σχέση με τους αποσπασμένους εργαζόμενους στη σχετική οδηγία. Συμφωνώ με όσα προελέχθησαν στην ακρόαση της Μάριαν Τάισεν ότι η Επιτροπή θα προβεί σε μια στοχοθετημένη αναθεώρηση της οδηγίας σε σχέση με τους αποσπασμένους για να αποφευθεί ο κίνδυνος του κοινωνικού ε, dumping και για να ορίσουμε έναν ελάχιστο μισθό στη χώρα υποδοχής. Εδώ υπάρχουν ορισμένα παραθυράκια τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να αποφύγουμε μία υπερβολική ερμηνεία. Άρα υποστηρίζω την πρωτοβουλία της ε, Μάριαν Τάισεν και θα την υποστηρίξω. Ως προς οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες ε, μου υποβλήθηκε η ερώτηση ήδη μία φορά και συμφωνώ με την πρόταση της Μαριαν Τάισεν και θα την ε, υποστηρίξω. Ε, ίσως να μην χρησιμοποίησα την ίδια διατύπωση με της Μαριαν Τάισεν, αλλά αυτό εννοούσα. Όσον αφορά το θέμα το οποίο θίξατε ε, σε σχέση με την τομεακή αυτή συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δυνάμει των Κοινωνικών Εταίρων έχει υποστηρίξει τη σχετική νομοθεσία και θα την προωθήσει. Επίσης, παράλληλα, λάβαμε ένα αίτημα από 10 κράτη-μέλη να μην προωθήσουμε αυτή την τομεακή ρύθμιση Και συνεπώς ε, η πρόταση αυτή γίνεται δεκτή σχεδόν ε, ομόφωνα. Έχει προταθεί σχεδόν ομόφωνα. Όταν λοιπόν προωθήσουμε αυτή την νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί, 10 δέκα κράτη-μέλη την έχουν απορρίψει, κράτη τα οποία δεν προβαίνουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Ότμαρ Κάρας από το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Κύριε υποψήφιε Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ για το ότι αναφερθήκατε και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το, πρέπει, για το ότι θα πρέπει να περάσουν στο κοινοτικό δίκαιο όλες αυτές οι κατασκευές ε, ανάγκης ε, συμπεριλαμβανομένης της ε, Τρόικας. Και βεβαίως ε, και εδώ πέρα ισχύουν και όλες οι κοινωνικές ελευθερίες και δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια περαιτέρω βήματα βλέπετε ότι χρειάζονται για την εμβάθυνση της ε, Θεωρείτε πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορούσε να γίνει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και θα μπορούσε ο υφιστάμενος μηχανισμός να αποτελέσει την βάση ενός διευρυμένου κοινωνικού διαλόγου. Okay, uh, thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρας. Αρκετές ε, ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω από τη μεσαία με το ε, μηχανισμό σταθερότητας και το αν θα γίνει Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ξέρουμε πως αρχικά υπήρχαν κάποιες συζητήσεις για κάτι τέτοιο, τελευταία δεν τις έχω ξανακούσει, οπότε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός σταθερότητα υπάρχει. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε ως μία μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα είναι να έρθει ο μηχανισμός εντός του κοινοτικού πλαισίου. Αυτή τη στιγμή είναι στο διακυβερνητικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να γίνει μία αλλαγή της συνθήκης για να μπει στο κοινοτικό πλαίσιο και νομίζω πως ε, και ως γενική προσέγγιση ε, το τόνισα αυτό πως πρέπει να συνεργαστούμε όσο γίνεται ε, στο κοινοτικό πλαίσιο και πολλά από αυτά τα διακυβερνητικά στοιχεία τα οποία δημιουργήσαμε νομίζω πρέπει να μπουν σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης για ζητήματα μακροοικονομικής διακυβέρνησης οπωσδήποτε είναι περίπλοκο το ζήτημα και έχουμε τώρα διαφορετικά επίπεδα μακροοικονομικής διακυβέρνησης και πρέπει να τα ενσωματώσουμε σε ένα ενιαίο και να έχουμε κάτι το συνολικό που θα είναι πιο εύκολα αντιληπτό, ένα γενικότερο πλαίσιο. Και Αυτό νομίζω θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της ε, αναθεώρησης των μακροοικονομικών πρακτικών μας και των συνομιλιών με τους κοινωνικούς εταίρους. Σας ευχαριστώ. Άκνες Χιουγγέριους από τους Σοσιαλδημοκράτες. Εδώ είμαι, ευχαριστώ. Θα κάνω την ερώτησή μου στα Ολλανδικά. Κύριε Ντομπρόφσκης μιλήσατε για μια κάποια ισορροπία της οικονομικής ε, και της κοινωνικής πολιτικής και αυτή είναι και η ερώτησή μου. Αυτό το θέμα αφορά. Γιατί τελευταία βλέπουμε πολλές αποφάσεις του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ε, που μιλάει για την οικονομική ελευθερία και το κόστος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και βλέπουμε μια τάση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό για την κατεύθυνση που έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μιλάμε για απαγόρευση αναγνώρισης ε, κατώτατου μισθού. Λέει πως κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους κανόνες της οικονομικής ε, ελευθερίας όταν μιλάμε για υπεργολαβία σε άλλο κράτος. Και βλέπουμε δηλαδή διάφορα φαινόμενα για τους αυτοαπασχολούμενους, για συμβόλαια που δεν αναφέρουν ώρες εργασίας κτλ. Το ερώτημά μου είναι ποια είναι η δική σας η προσέγγιση, τι θα κάνετε ε, για να αμβληνθεί αυτή η ένταση μεταξύ θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων αφενός και οικονομικών ελευθεριών από την άλλη. Τι θα κάνετε για να υπάρξει ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Πέτροπο. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, για τις εξελίξεις ε, στην αγορά εργασίας βλέπουμε πόσο τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες ε, υπάρχει μια αγορά εργασίας ε, δύο κατηγοριών. Υπάρχουν κάποιες νέες ιδέες ε, με αυτά τα συμβόλαια μηδενικών ορών ή ψεύτο αυτοαπασχολούμενους ε, για να παρακαμφθεί η νομοθεσία. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε μαζί με τα κράτη-μέλη ακριβώς ε, για να βελτιωθεί και η ευελιξία με ασφάλεια όπως λέγεται αλλά ταυτόχρονα να δούμε και τα διάφορα παραθυράκια τα οποία χρησιμοποιούνται για να, αποφευχθεί, για να παρακαμφθεί η νομοθεσία της αγοράς. Αυτό το πρόβλημα πράγματι με τους ε, υποτίθεται ελεύθερους επαγγελματίες ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται. Ακριβώς για να δούμε πώς θα γίνουν πιο ομοιόμορφες ε, οι αγορές εργασίας και να μην έχουμε αγορά εργασίας δύο κατηγοριών με κάποιους να προστατεύονται και κάποιους άλλους όχι. Όσον αφορά τώρα τις αποφάσεις του δικαστηρίου, ξέρετε πως ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα σχολιάσω και δεν θα αφισβητήσω τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου. Το εμείς απλά τις εφαρμόζουμε και βεβαίως ε, ε, κοιτάμε ταυτόχρονα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Η Ιβάνα Μάλετιτς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκη, σε χαίρομαι διότι είσαστε υποψήφιος για την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ε, πολιτική με συγχωρείτε έχετε τις κατάλληλες γνώσεις και πείρα ως πρώην Πρωθυπουργός και δείξατε ότι έχετε θάρρος και είσαστε αποφασισμένος. Πολλοί εμπειρογνώμονές σας συνεργάστηκαν με την Κροατία σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η συνεργασία σας. Είχατε μεγάλη πείρα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ορίζετε την πολιτική συνοχής και τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Πώς μπορείτε να επιλύσετε θέματα πληρωμών από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό στα κράτη-μέλη, διότι αυτό είναι ένα από τα βασικά προσκόμματα στην ανάπτυξη και την απασχόληση απάντηση. Ως προς την καλύτερη συνδεσιμότητα χωρών και συστάσεις για την πολιτική συνοχής. Αυτό το θέμα προωθείται τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται τις ε, εταιρικές συμφωνίες και τα ε, επιχειρησιακά τους προγράμματα με την Επιτροπή και μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής είναι ε, η χρηματοδότηση προγραμμάτων συνοχής να ακολουθεί συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και να έχει μια συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Δηλαδή καλύτερη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, δηλαδή περισσότερο να δούμε το κοινωνικό σκέλος, την κοινωνική πτυχή. Για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τα κοινωνικά προβλήματα των ε, χωρών. Ως προς τις πληρωμές, αυτό το θέμα δεν άπτεται του χαρτοφυλακίου μου. Αφορά το χαρτοφυλάκιο της Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Έχουμε όμως με ένα θέμα του Συμβουλίου το οποίο μπλοκάρει τις ε, πληρωμές και ξαναμπαίνει στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές που ορίζει σε κατώτερο επίπεδο από αυτό που έχει οριστεί από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επειδή πρόκειται για διαθεσμική συμφωνία, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε το Συμβούλιο να σεβαστεί αυτή τη διαθεσμική συμφωνία και να μην δημιουργεί τέτοιες κρίσεις με τις πληρωμές. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Χαβιέ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες έχετε το λόγο. Καλό σας απόγευμα. Όπως ε, γνωρίζετε, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν από την Τρόικα οδήγησαν σε δρακόντριες ε, περικοπές και καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες. Υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη τέσσερα χρόνια πριν και επίσης υπάρχουν και αντιπαραγωγικά μέτρα με συγκεκριμένες ελλείψεις, με συγκεκριμένο δημοκρατικό έλλειμμα. Ο πρόεδρος Γιούνκερ κατά την ορκομοσία του ε, είπε ότι θα ε, αναθεωρήσει αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα σχέδια κοινωνικής αποτίμησης πώς ορίζονται Επίσης μπορείτε να μας πείτε ότι αυτά, αυτές οι εκτιμήσεις, οι αξιολογήσεις μάλλον δεν θα μείνουν επί χάρτου. Επίσης, εάν υπάρχει μία αξιολόγηση που θα δείξει αρνητικό αντίκτυπο, θα, αντίκτυπο, θα την αποσύρετε ναι ή όχι. απάντηση. Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης συζητήσαμε επί μακρόν το θέμα των θέσεών μας όταν ε, ε, αναδυθήκαμε από την κρίση και συζητήσαμε και τα μέτρα της ε, Τρόικας και στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών επιπτώσεων. Στόχος της νέας Επιτροπής είναι να διορθώσει τα μέτρα αυτά και να λάβει αποφάσεις λαμβάνοντα υπόψη όχι μόνο την δημοσιονομική βιωσιμότητα αλλά και διενεργώντας ε, μελέτες αντικτύπου, κοινωνικού αντικτύπου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής και η κυρία Τάισεν που θα είναι υπεύθυνη για κοινωνικές υποθέσεις, για τις κοινωνικές υποθέσεις, θα ασχοληθούν με αυτή την πτυχή του θέματος και εγώ θα συνεργαστώ ε, έτσι ώστε αυτή η δέσμευση να μην παραμείνει επί χάρτου. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάινς Μπέκε από το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκης ως αστεργακός και μέλος ε, της Επιτροπής Κοινωνικών και Απασχόλησης χαιρετίζω αυτά τα οποία είπατε για τον κοινωνικό διάλογο και τον ρόλο που θα πρέπει να έχουν οι κοινωνικοί εταιροί στο μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά πάρα πολλά προβλήματα νομίζω οφείλονται στην ε, πολιτική των κρατών μελών λόγω και της επικουρικότητας. Θα μπορούσατε να ε, μας περιγράψετε έναν μηχανισμό για να διδάσκονται κάποιες χώρες από αυτά τα οποία έχουν εφαρμοστεί επιτυχημένα σε άλλες χώρες μέλη. Και πώς θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε δεσμευτικούς κανόνες για ε, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Νομίζω το κάνατε, το κάνατε αυτό στη χώρα σας. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Όσον αφορά την επικουρικότητα, είναι σαφές πως είναι μια βασική αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή μόνο τα ζητήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζονται καλύτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν σαφώς ε, ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία ε, θα λύνονται σε αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι η αρχή και την εφαρμόζουμε. Όσον αφορά τώρα την ανταλλαγή βέλτιστων ε, πρακτικών και την εμπειρία άλλων κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει η ε, Κομισιόν και στον τομέα επίσης της ε, κατάρτισης και των της ε, διαβίου εκπαίδευση, νομίζω πως μπορούμε να δούμε το γερμανικό σύστημα της ε, μαθητείας, αλλά και άλλα συστήματα που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη για να διδαχτούμε από αυτά. Γιατί ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην αγορά εργασία είναι πως δεν ανταποκρίνονται τα προσόντα των νέων όπως βγαίνουν από το σύστημα εκπαίδευσης σε αυτά τα οποία απαιτεί η αγορά εργασίας. Οπότε πρέπει πραγματικά να δούμε καλύτερη διασύνδεση ε, μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων. Γεώργη Πυρίνσκι από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, η οδηγία για τις ε, μονοπρόσωπες ΕΠΕ σαφώς ε, δεν δίνει καμία εγγύηση για τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση, την διαβούλευση και τη συμμετοχή στο ΔΣ. Οπωσδήποτε, όταν μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση, ε, αναλαμβάνετε εσείς το να αποσύρετε αυτό το σχέδιο οδηγίας και να καταλήξετε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς το πολύ επικίνδυνο αυτό παραθυράκι στο σχέδιο οδηγίας θα κλείσει και θα ξεκινήσετε διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και δεσμεύστε να μην ξαναφέρετε τέτοια πρόταση χωρίς ε, πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση για την βασική, τις βασικές αρχές της νέας ε, Κομισιόν ε, ήδη αναφέρθηκαν είναι δηλαδή να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ ε, της οικονομικής και της κοινωνικής διάστασης για να διασφαλίσουμε την προστασία μεταξύ άλλων των εργαζομένων. Τώρα θα με συγχωρήσετε, δεν μπορώ να πω κάτι για τη συγκεκριμένη οδηγία, αλλά ευχαρίστως να το δω το ζήτημα και να με ενημερώσει και η αρμόδια υποψήφια επίτροπος, η κυρία Τάισεν, και εάν α, υπάρχουν κάποια παραθυράκια όπως είπατε, Νομίζω πως η Κομισιόν θα τα κλείσει ή θα αποσύρει αυτή την ε, τροπολογία. Γνωρίζουμε πως ο υποψήφιος πρόεδρος, ο κύριος Γιούνκερ, δήλωσε πως ε, υπάρχει κάποια δυνατότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Refit για καλύτερη, καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο να υπάρξει απόσυρση πολλών ε, νομοθετικών προτάσεων και οπωσδήποτε θα κοιτάξουμε και αυτήν. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή για αυτή την οδηγία. Αλλά μαζί με την ε, κυρία Τάισεν ε, ευχαρίστως να το εξετάσουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα σας στείλω κάποια απάντηση αργότερα διμερώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παρβάνοβα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ σε υποψηφίο αντιπρόεδρο. Ήρθαμε σε επαφή πολλές φορές σε διασκέψεις κορυφής του ΕΛΚ, όπου ε, δείξατε τις μεταρρυθμίσεις, καταδείξατε ότι ε, έγινε και υπήρξε πρόοδος στη χώρα σας, επειδή ακριβώς κάνατε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις, τις βουλευτικές χτεσινές εκλογές. Η το κόμμα μου ε, μπόρεσε να επικρατήσει έναντι των αντίπαλων κομμάτων. Άρα θα ήθελα να μιλήσω για ένα βασικό θέμα. Η απειλή μιας Ευρώπης δύο ταχύτητων αποτελεί δαμόκλειο σπάθη ιδιαίτερα για τις ε, χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης ή αποσκοπούν σε αυτό. Πώς μπορείτε να μας ε, εγγυηθείτε ότι η Ευρωζώνη δεν θα υποβαθμίσει τις άλλες ε, χώρες μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης απόφασης για τις οικονομίες των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Στα εισαγωγικά μου σχόλια σας μίλησα για την εξής ανάγκη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανελιχθεί σε επίπεδο των 28 κρατών. Επίσης η Ευρωζώνη θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή σε νέα δηλαδή να προσχωρήσουν αν το επιθυμούν και θα πρέπει η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά σε επίπεδο 28 κρατών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολιτικές και ζητήματα που φύγουν την Ευρωζώνη, διότι οι χώρες αυτές μοιράζονται το ίδιο νόμισμα. Όμως η Ευρωζώνη δεν θα πρέπει να γίνει, να μετατραπεί σε μία αποκλειστική ζώνη μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Άρα οι αποφάσεις σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο 28 κρατών μελών και θα αρκεστώ σε αυτή την αρχή ως νέος επίτροπος. Η Μαρία Χαουρετήκης από τις Σοσιαλιστές. Κύριε Ντομπρόφσκης, αν πραγματικά θέλετε να αποσοβηθεί η κρίση, θα πρέπει να μεταθέσουμε τις προτεραιότητές μας και για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να επιδοθούμε σε επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι δημοσιονομική ενοποίηση. Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο προτεραιότητες, επενδύσεις ε, και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μέσα στα πλαίσια των συστάσεων προς τις χώρες μπορείτε να μας πείτε στην ετήσια ε, μελέτη πώς θα λάβετε υπόψη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να υπηρετήσει αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ερώτηση, την επερώτηση. Και όπως ε, αναφέρθηκα και στις ε, αρχικές μου δηλώσεις, η προτεραιότητα της νέας Επιτροπής είναι επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση. Εδώ θα εστιάσουμε την προσοχή μας και στα πλαίσια της ε, νέας ενιαίας ετήσιας πορείας μας, όπως ε, τόνισε και ο πρόεδρος Juncker. Ε, Τώρα, ως προς την ευελιξία μέσα στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας, ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η, ρύθμιση και ιδιαίτερα για τις ε, χώρες που έχουν ρυθμό ανάπτυξης ε, κάτω από το 0 ή μείον 4% θα πρέπει να απαλλαχθούν από αυτές τις υποχρεώσεις, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μείον 1,5% με μείον 4% που σημαίνει είτε μη προσαρμογή ή μη δυνατότητα προσαρμογής. Ε, επίσης ε, υπάρχουν και ρήτρες διασφάλισης ιδιαίτερα όταν έχουμε συγκεκριμένα ε, δημοσιονομικά αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ρήτρα εξαίρεσης και σε αυτή την ε, περίπτωση γίνεται προσαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Υπάρχουν και άλλοι τομείς ευελιξίας, όμως ε, εντάσσεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα κράτη-μέλη ομοιογενώς. Ο κύριος Λάγκερ, που είναι ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης. Νομίζω έχετε αποδείξει μέσα από αυτά τα οποία κάνατε στη χώρα σας πως μπορείτε να πείσετε μεταρρυθμίσεις και οικονομία. Αυτά τα οποία προτείνονται τώρα, ευρωομόλογα, περαιτέρω χρέος και αυτό το οποίο ακούμε να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός σταθερότητας για επενδύσεις είναι συνταγές ε, που είναι μεν υποσχέσεις αλλά δεν βοηθάνε σε τίποτα. Έχω το ίδιο ερώτημα που έκανε στον κύριο Μοσκοβησή για εσάς. Τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση, γιατί γι' αυτό ακριβώς είναι οι κανόνες. Σύμφωνα με το άρθρο 6, Μοσκοβησή και Ντομπρόφσκης θα πρέπει να διαμορφώνουν τους κανόνες από κοινού. Επίσης, για την αποχώρηση από την Ευρωζώνη. Πράγματι πρέπει να αλλάξει η συνθήκη, αλλά ε, τα κράτη, ε, κράτος, παραδείγματος χάρη μέλος, πρέπει να κάνει και ε, κράτος μέλος Ευρωζώνης, πρέπει να γίνει και η Σουηδία που εκπληρώνει τις συνθήκες, αλλά αρνείται. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις όπου είναι σαφή η συνθήκη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ήταν δύο νομίζω. Πρώτα απ' όλα τα... μία αφορούσε τον καταμπερισμό εργασίας μεταξύ μου και του κυρίου Μοσκόβηση. Οπωσδήποτε θα εργαστούμε ως ομάδα, θα συνεργαστούμε στενά και εγώ θεωρώ πως ο ρόλος μου είναι συντονιστικός και όχι ρόλος επόπτη ή κάποιος ο οποίος ε, θα προσπαθεί να διαχειριστεί ε, όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε συνεργασία με τον κύριο Μοσκοβησή σε διάφορες πτυχές και στην εξωτερική εκπροσώπηση και στο θέμα του να κάνουμε προτάσεις από κοινού. Και βεβαίως ο Επίτροπος κάνει την δουλειά του, αλλά υπάρχει η δυνατότητα και του Αντιπροέδρου της Κομισιόν να συνεισφέρει νωρίς την διαδικασία για να μπορούμε να πούμε πως είναι μια κοινή πρόταση. Συμφωνήσαμε νομίζω σε αυτό ως βασική αρχή και αυτή τη στιγμή οι ομάδες μας εργάζονται προς κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. θα είναι αυτό νομίζω τις ε, πρώτες εβδομάδες ούτως ή άλλως της νέας εντολής. Τώρα όσον αφορά τις χώρες εκτός Ευρωζώνης και τη Σουηδία γνωρίζουμε την κατάσταση, γνωρίζουμε τα αρνητικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και βεβαίως γνωρίζουμε το τι προβλέπει η συνθήκη. Αλλά σαφώς η Κομισιόν δεν μπορεί να αναγκάσει κάποια χώρα να μπει στο ευρώ. Νομίζω λοιπόν πως η Ευρωζώνη πρέπει να είναι ανοιχτή, διαδεθειμένη να δεχτεί νέα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορούμε να ε, βάλουμε κάποιον με το ζόρι. Ως Σουηδέζα θα μπορούσα να πω ένα ε, επιπρόσθετο ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και σας ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης για τις απαντήσεις σας. Τώρα έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για ε, μια καταληκτική δήλωση. Πέντε λεπτά πριν λήξει και η συνεδρίασή μας. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. So, uh, uh, Αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ευκαιρία, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τον μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που με υποβάλλατε που και που καταλαβαίνω θα απαιτήσουν περαιτέρω δουλειά και παρακολούθηση. Πάντως είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ στενά με το Ευρωκοινοβούλιο καθώς και εγώ ίδιος έχω διατελέσει ευρωβουλευτής για να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι σας οφείλω μια, μια απάντηση για μια ερώτηση που τέθηκε και με επικρίνατε που δεν μπόρεσα μέσα σε δύο λεπτά να την απαντήσω και αφορούσε τα σφάλματα τα οποία έγιναν στην Λετωνία ε, κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της κρίσης και νομίζω πως μπορείτε να βρείτε κάποιες απαντήσεις στις ειδικές συστάσεις προς τη Λετωνία. Υπάρχουν διάφορες συστάσεις πολιτικής όσον αφορά την ενίσχυση της ανεξαρτησίας μας στην ενέργεια. Πολύ σημαντικό θέμα σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο. Στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στα εισοδήματα συμπεριλαμβανομένων ε, των αλλαγών ε, στη συνεφορολογική πολιτική, ενίσχυση του δικαστικού σώματος, αντιμετώπιση προβλημάτων αφαιρεγγιότητας, Διάφορες λοιπόν συστάσεις ε, για τη χώρα μας που λάβαμε και που ε, εντόπισαν προβλήματα τα οποία θα έπρεπε η Λετωνία να αντιμετωπίσει. Ελπίζω πως η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί τώρα, γιατί πριν δύο μέρες μόλις κάναμε, είχαμε εκλογές, ε, Ελπίζω λοιπόν ότι θα δεχτεί και θα λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις συστάσεις η νέα κυβέρνηση και θα μπορέσει έτσι να αντιμετωπίσει τις πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Λετωνία. Όσον αφορά την εργασία της Νέας Επιτροπής, θα πρέπει και να τονίσω για μια ακόμη φορά πως πρόκειται για μια νέα δομή, οπότε δεν έχουν όλα ε, κουρδιστεί στην τελευταία λεπτομέρεια, αλλά μπορώ σαφώς να σας πω ότι όλοι οι υποψήφοι επίτροποι με τους οποίους έχω συνομιλήσει διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, είναι πρόθυμοι για να εργαστούν ομαδικά, ε, οφείλω μου τους ή άλλως να δουλέψουμε ομαδικά ακόμα και αν ε, προερχόμαστε από διαφορετικά πολιτικά ε, κόμματα, ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να αποδώσουμε ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα θέματα που ανησυχούν τον κόσμο. Τα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης, τα θέματα της απασχόλησης, της εξέλιξης των μισθών, τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για αυτή την ακρόαση και πραγματικά προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί σας και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Just a few remarks on the... Μερικές παρατηρήσει για την διαδικασία που θα ακολουθήσει. Θα γίνει κοινή αξιολόγηση, συνεδρίαση αξιολόγηση με τους Προέδρους των δύο Επιτροπών και τους συντονιστέ. Θα γίνει στις 7 ε, απόψε στην αίθουσα 3G2 στο κτίριο ASP θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη τις διάφορες ε, ανησυχίες ε, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ε, επιστολής αξιολόγησης και που θα κυκλοφορήσει αργότερα απόψε. Η προθεσμία για σχόλια για την επιστολή είναι πρωινή, αύριο στις 7 Οκτωβρίου δηλαδή και οι συντονιστές είναι οι, άνθρωποι επαφής και ζητώ από τους συντονιστές ε, της Επιτροπής Απασχόλησης να έρθουν εδώ κοντά μου για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε τώρα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Οι συντονιστές λοιπόν ε, της Επιτροπής Απασχόλησης παρακαλώ ελάτε εδώ κοντά μου στο Προεδρείο. Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά κύριε Ντομπρόφσκης ευχαριστώ όλα τα μέλη των δύο Επιτροπών που ήσασταν σήμερα εδώ και που θέσατε ε, ευφυείς ερωτήσεις.